να ξεκινήσουμε για με την ψηφοφορία για τι κλινικέ δοκιμέ φαρμάκων. Στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξη. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έχετε όλε τι κάρτε σα μαζί. Genau, deswegen. Ja, aufmachen. Bitte. Clinical Trials. So. Hat jeder... Κλινικές δοκιμές φαρμάκων. Έχετε όλες τις κάρτες σας, τις κάρτες ψηφοφορίας. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, κανένας κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Και συνεχίζουμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση Μπελιέ. Η κυρία Μπελιέ θέλει να προβεί σε μια δήλωση σχετικά. Καλό θα ήταν να έχει καταστάσει, βέβαια, η συγγήτρια. Στην περίπτωση αυτή, να κοιτάξουμε το θέμα του καπνού. Να προχωρήσουμε στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης, αφού λείπει η συνάδελφος για τον καπνό. Προϊόντα καπνού. Εδώ θα επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Έναξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. E Από το ECR περισσεύει μία ψήφος. Από το ECR παρακαλώ περισσεύει μία ψήφος. Να συμφωνήσουμε αν θέλετε. Από το ECR είσαστε υπεράριθμοι. Έχετε μία ψήφο παραπάνω.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 So, vielleicht kann bitte ein Technik. Αν θα θέλετε κάποιος από τους τεχνικούς να μας βοηθήσει. Wir müssen die θα πρέπει να προγραμματίσουμε, να αναπρογραμματίσουμε τις ε, συσκευές ψηφοφορίας από Επιτροπή Απασχόλησης σε Επιτροπή Περιβάλλοντος. Γι' αυτό λοιπόν λάθος έκανα που είπα και άδικο είχα που είπα ότι ε, είναι ένας υπεράριθμος από το ECR. Hi. So, wir sind jetzt hier in 4Q2 im Envy-Mode und wir können jetzt... Μάλιστα. Έτοιμοι είμαστε και τώρα μπορούμε να περάσουμε πάλι στην έκθεση Μπελιέ, να συνεχίσουμε κανονικά με την ημερησία διάταξη στο 9, όπως είπα, τη ημερησίας διάταξη. Η κυρία Μπελιέ θέλει να κάνει μια δήλωση ή μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν. Merci, Monsieur le Président. Une, une minute. Ένα λεπτό μόνο σχετικά με την συγκεκριμένη ψηφοφορία. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ δύσκολες. Θα υποστηρίξω ότι πάρα πολλές χώρες ήταν εναντίον της κοινοτικής μεθόδου και των νέων κανονισμών στον τομέα της βιοπικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστέρησε χαρακτηριστικά να μας υποστηρίξει. Η Λιθουανική Προεδρία μας περιφρόνησε σαν κοινοβούλιο. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης δεν είναι τόσο φιλόδοξο όσο θα το επιθυμούσα και οι θέσεις τις οποίες ε, κατέληξε το Κοινοβούλιο από το 2013 μας επιτρέπουν να έχουμε ένα κανονισμό που θα μπορέσει να καταστήσει ικανή την Ένωση να επικυρώσει την Αγκόγια και να πάρει μέρος και στο, στην διάσκεψη του ΟΗΕ στην Κορέα στο τέλος του χρόνου. Ατέλεστο πλαίσιο, αλλά τουλάχιστον καταπολεμούμε τη βιοπειρατεία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις για την βοήθειά τους και να θυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα είμαστε απαιτητικοί από την Επιτροπή σχετικά με τις εκτελεκτικές πράξεις του άρθρου 17 της Ναγκόγια και, ε, και του άρθρου 7 του κανονισμού μας. Μάλιστα να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία, μία λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας και αν ψηφίσατε όλοι, πέρας της ψηφοφορίας. 51 ψήφοι υπέρ, τρει αποχές, εγκρίθηκε λοιπόν και περνάμε τώρα στο 10 τη ημερήσιας διάταξης. Κατευθείαν στην ψηφοφορία περνάμε. Ο Chris Τέιβις. Πρόεδρε, νομίζω ότι η έκβαση των τριμερών διαλόγων ήταν εξαιρετική και οι διαπραγματευτές έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά το άρθρο 18 που αφορά τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα ξαναδιατυπώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και υπάρχουν πάρα πολλές αβεβαιότητες και συγχύσεις στο κείμενο και δεν μας εκπλήσει αυτό κάτω από τις συνθήκες ε, τις οποίες προετοιμάστηκε το κείμενο. Θα περάσει η πρόταση βέβαια και θα πάμε στην Ολομέλεια, αλλά εμείς θέλουμε να τηρήσουμε επιφυληκτική ε, στάση για να δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή πριν την Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ, Chris Davis. Ε, μπορούμε λοιπόν να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία και αν ψηφίσατε, συγγνώμη, αν έχετε βάλει όλη τη κάρτα σας, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Με 49 ψήφους υπέρ 7 κατά 4 αποχές επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα της τριμερούς διαλόγου. Συγχαρητήρια στη Λίντα Μακέδων. Dann geht's, dann geht's weiter. Συνεχίζουμε λοιπόν στο σημείο 8 που το συζητήσαμε σήμερα λέει ο πρόεδρος στο 11 της ημερήσιας διάταξης ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε στο 11 στο 11 Αν ψηφίσατε όλοι Α, ξέρετε, είναι κάποιος υπεράριθμος από τους σοσιαλδημοκράτες. Ψηφίσατε όλοι, πέρα της ψηφοφορίας. 34 ψήφοι υπέρ, 21 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα λοιπόν θα περάσει στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο, όπου θα γίνει και η εξέταση. Συνεχίζουμε με την ψηφοφορία για την έκθεση του Bart Stas. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 10, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 69 με προφορική τροπολογία από πλευράς, ε, για μένα στη σελίδα 5. Η 69 με προφορική τροπολογία. Το βρήκατε στη σελίδα 5 στο δικό μου κατάλογο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στην 21 περνάμε τώρα στην επόμενη σελίδα. Υπέρ του εισηγητή. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε τώρα στην 24 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Consolidated 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε στην 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Από την 28 και την 31 μαζί παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 2. Υπέρ. Κατά. Α, εγκρίνεται η 35. Κατά. Αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3 και η 37 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 39. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται με σαφή διαφορά η 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται η 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ. Κατά. Α, εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συνεχίζουμε στην 46 υπέρ. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη 3 ε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία, καταρχάς ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Τώρα μάλιστα, εντάξει. Πέρασε ψηφοφορία. 59 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 0 αποχές. Και τώρα περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Αν ψήφισετε όλοι, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. 54 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. Εγκρίνεται τώρα να ζητήσω από τον ε, εισηγητή κατά πόσον θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα και τους κοιόδους εισηγητές, αλλά να ευχαριστήσω και όλους τους ε, συναδέλφους ε, που κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ακολούθησαν τη γραμμή των σκιωδών και του εισηγητή. Θα ήθελα να σας ζητήσω εντολή για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο στα πλαίσια τριμερούς διαλόγου να ξεκινήσουν και ελπίζουμε μήπως και μέχρι τα τέλη της θετίας να καταφέρουμε να καταστήλξουμε σε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Μάλιστα, θέλει λοιπόν και ζητά εντολή ο εισηγητής. Θέλουμε 36 ψήφους υπέρ για να δοθεί η εντολή στον εισηγητή. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ, είναι Αν ψηφίσετε όλοι. Τρεις ψήφοι λοιπόν. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. 60 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια Μπαρτ και ευχόμαι να πάνε καλά διαπραγματεύσεις. Jetzt geht's weiter. Να συνεχίσουμε με την υγεία των ζώων. hier Ja. Mhm. Und zwar mit 190 dafür. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να ψηφίσουμε παρακαλώ για την 230 ηλεκτρονικά. Και αν ψηφίσατε όλοι, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Έγκρινεται. Να περάσουμε στην ενοποιημένη 7. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την ενοποιημένη 7. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι παρακαλώ. Πέρασε. Έγκρινεται. Και τώρα συνεχίζουμε στο δεύτερο τμήμα της αναποιημένης της 34. Ε, το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Στη 43, τέσσερα τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ενοποιημένη 4 υπέρ. Consolidated 4. Ενοποιημένη 4. Στην επόμενη σελίδα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τη 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 47. Έναρξη και πέρας ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 34 κατά. Αν 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία νομίζω διαμορφώνεται, αλλά αν το ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν είμαι σίγουρος. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 48. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Η 236 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Και περνάμε τώρα στην 239 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 241 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 242 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 243 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 244 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 245 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 246 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ. Το 246 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Ε, περισσεύει ένα από του σοσιαλδημοκράτε όμω. Τώρα εντάξει. Απορρίπτεται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 248 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα για την 250 παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 54. Υπέρ. Α, καταπίπτει. Καταπίπτει. Η 59. Μαζί με την 60, την 64. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε στην ενοποιημένη Συγγνώμη. Με την 61 δεύτερο τμήμα. 61 δεύτερο τμήμα ψηφίσουμε, παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Δεν ε, φαίνεται σαφώς να ψηφίσουμε την 61 ηλεκτρονικά παρακάτω. Δεύτερο τμήμα. Αν ψήφισατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και συνεχίζουμε στην ενοποιημένη 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές και πάλι το αποτέλεσμα είναι Το αποτέλεσμα γι' αυτό το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορίας παρακαλώ. Για την ενοποιημένη 6. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 254 υπέρ. Μαζί με τη 255 και τη 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ζητείτε έλεγχο για την 254, 255, 256 από κοινού. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, αν ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε με τη 257 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 81 και η 82 από κοινού παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 81 και 82 παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την 263 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 84-85 μαζί παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία για την 84 και 85. Αν ψηφίσατε λοιπόν όλοι, ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο σημείο αυτό. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα από κοινού την 86, 87, 88 και την 90. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 266 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 267 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 268 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 269 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Για την 268. Εγκρίθηκε είπατε. Εγκρίθηκε λέει ο πρόεδρος. Okay, 200. Για την 268 παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Mm. Πέρα ψηφοφορίας. Αγαπητέ Καρλ Σλούτερ, ήταν πιο πολύ πράσινη από ότι η κόκκινη, άρα εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ε, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 94 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας και αν ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Άποχες. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα, παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι, πέρας ψηφορίας. Σαφώς εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 98. Ψήφισατε όλοι. Πέρα του ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν. Η επόμενη καταπίπτη 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 272 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 273 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 101 και αν ψήφισατε όλοι. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 102 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 105. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 275 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111, 112 και 113 unblock παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. 115. Μάλιστα. 115 λοιπόν υπέρ. 115 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 277 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 καταπίπτει. Και περνάμε λοιπόν Συνεχίζουμε στην 125-124. Ε, ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 127 Την 127 παρακαλώ ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 133 ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 286 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 288 απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 288. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε τώρα στην 291 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 292 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 293 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 295 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 296 υπέρ κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 296. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Περισσεύει πάλι ένας από τους σοσιαλδημοκράτες. Πέρασε. Α, απορρίπτεται. 297 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 298 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 299 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 300 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 301 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται, εγκρίνεται συγγνώμη η 302 διευθυντή πρόεδρος εγκρίνεται η 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 304. Ψήφισετε όλοι παρακαλώ. Την 304. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 305 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 309 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Την 309 λοιπόν την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισατε παρακαλώ όλοι. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται. Την 310 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Την 142 λοιπόν την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 313, 314 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 315 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 316 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 317 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 147 είναι προσθήκη 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 318 υπέρ όχι καταπίπτει 319 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 421 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι ξεκάθαρο. Παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία 321 άρχεται, ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται. Η 322 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 323, ε, 324 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 155. Καταπίπτει. Όχι. Όχι, πρέπει να ψηφίσουμε για την 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 327 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 331 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 3.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά πηγαίνουμε κάποιες τροπολογίες και συνεχίζουμε με την 3.44 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 3.55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για την 165 αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ναι, εγκρίθηκε. 358 υπέρ. Κατά. Ξανά. 358 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Συγκρίνεται. 359 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 361 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 360 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα 369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 371 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 372 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.73 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 3.74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.77 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 3,78 ειπε κατά αποχές, απορρίφθηκε. 3,79 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 3,80 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 172 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίθηκε 173 υπέρ, κατά αποχές, δεν είναι ξεκάθαρο. 173 ηλεκτρονική επαλήθευση. αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε ναι. να. 381 υπέρ. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Ε, έτρεχα πολύ. Είναι 173 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται πέρας τα ίδια βγήκαν ε, 389 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 382 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 175 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 383 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 384 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο 34 ηλεκτρονική ψηφοφορία προσοχή ψηφίζουμε ηλεκτρονικά μην ξαναγίνουν τα ίδια πέρας εγκρίθηκε να 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 386 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 387 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 179. Παρακαλώ, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται όντως. 180 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 388 υπέρ. Κατά. Απόχε. δεν είναι ξεκάθαρο ηλεκτρονική επαλήθευση για την 388. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 184. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται και τώρα συμβαστική 1. ειπε Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 185 είπε Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 189. Είπε. Κατά. Απόχες. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ψηφίζουν ηλεκτρονικά για τα 189. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Καταπίπτει. Μάλιστα. Καταπίπτει ή δεν καταπίπτει. Ένα λεπτάκι. Καταπίπτει. Δεν χρειαζόταν να την ψηφίσουμε. 192 ε, υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 202 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο. 202 ηλεκτρονική επαλήθευση. Εψήφισαν όλοι. Ε, πέρας. Εγκρίθηκε τελικά. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 205. Όχι. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 213 κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 216 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 όχι καταπίπτει 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροπολογία 1 σχετίζεται με τη 218 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται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 κατά αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα 229 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα το ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε Συγχαρητήρια στην Καρτίκα Λεωτάρ. Και τώρα συνεχίζουμε. Να συνεχίσουμε στο 14 της ημερήσιας διάταξης. Τροπολογία 84, υπέρ. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 19 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές να επαληθεύσουμε την 19 παρακαλώ ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με την 108 υπέρ. Κατά. Άποχες. Την 108 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 καταπίπτει, 23 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 117 ή 118 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Άλλη μια φορά, αν θέλετε, την 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Ζητείτε έλεγχος για την 119. Παρακαλώ, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 119. Αν ψήφισετε όλοι, πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται με σαφή διαφορά. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ψηφίσουμε και αυτή ηλεκτρονικά παρακαλώ. Την 120 την ελέγχουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε, καταπίπτουν οι επόμενες. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. πίπτη η 125. Υπέρ. 32 Παρακαλώ ψηφίζουμε την 32. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126. Α, συγγνώμη. 120... 134. Η 34, συγγνώμη. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα να ψηφίσουμε την 130 μέχρι την 139 μπλοκ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 130 μέχρι 139. Από κοινού και ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφέ. Για την 141 παρακαλώ, ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, αν ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143 καταπίπτει. 144 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ε, ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα ψηφορίας. Ψήφισατε όλοι. Τώρα, τώρα ολοκληρώνεται. Γιατί περισσεύει ένας από τους σοσιαλδημοκράτες, παρακαλώ. Περισσεύει ένας από τους σοσιαλδημοκράτες. Είστε υπεραριθμοί. Εντάξει. Τώρα εντάξει. Εγκρίνεται. 146 καταπίπτει. Η 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 5 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μόνο 10 συνάδελφοι ψήφισαν. 45 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Ηλεκτρονικά ας ψηφίσουμε την 155. Ψηφίσατε όλοι. Την 45. Την 45 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ. Εάν ψηφίσατε όλοι. ολοκληρώνω την ψηφοφορία. Μάλιστα, εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ενωπημένη 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ.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 Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να ψηφίσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 173. Ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. 52 υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3 να ψηφίσουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ. Να την ελέγξουμε παρακαλώ. Την 78. Την 78 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 9 στο πρώτο τμήμα, τη 9, επειδή εγκρίθηκε η 60. Και τα δύο τμήματα αυτά ψηφίσουμε. Πρώτο τμήμα της 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη τη ψηφοφορία. Ψήφισετε όλοι. Πέρας. Συγχαρητήρια. Κύριε Ρώση. Μπράβο σας. 58 ψήφοι υπέρ. 6 αποχές, 0 ψήφοι κατά. Και έτσι λοιπόν περνάμε στην έκθεση Haug για την απαλλαγή να σας πω ότι έχω ήδη κάποια νοσταλγία γιατί θα είναι η τελευταία απαλλαγή που ψηφίζουμε με την κυρία Χάουκου τουλάχιστον στον τρέχουσα θητεία με αυτό το κοινοβούλιο. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 1 και 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 και 4 ταυτόσημες. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 6 και η 7 με προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα. Πρώτα με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με την 8 και την 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 10 και 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 12 και 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 14 υπέρ. Α, θέλετε να ελέγξουμε την 12 και την 13, μάλιστα. Να ψηφίσουμε λοιπόν μαζί ηλεκτρονικά την 12 και την 13. Ψηφίσετε παρακαλώ όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. 39 ψήφι υπέρ, 25 κατά εγκρίνεται. 14 στη συνέχεια υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 14. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 την ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 16. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει, η 17 και η 18. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ελληνικά. Ανάξη ψηφοφορίας. Πέρας. Υπεράριθμος ένας από τους δημοκράτες. Πέρας. 56 υπέρ, 7 κατά, 0 αποχές. Και συνεχίζουμε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Τροπολογία 1 λέει ο Πρόεδρος. Κατά, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 2 και οι 3 μαζί, ταυτόσιμες. Ψηφίσονται από κοινού. οι δύο και οι τρία θα ψηφιστούν μαζί με προφορική τροπολογία. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Ναι. Στο 16 είμαστε. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. So, wir werden es ja wohl die intellektuelle Leistung hinbekommen. Europäische Medizin Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 και 3 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 και 7 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 και 9. Ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ηλεκτρονική ψηφορία. Έναρξη. Πέρας. 56 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, 0 αποχέ. Συγχαρητήρια για το Χάγκο. επόμενη αρχή από τη Φιλανδία. Ξέρετε τι εννοώ. Χημεία, χημική. Ευρωπαϊκό οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην αρρύθμιση. Η γραμματεία ζητά συγγνώμη Μιλάμε τώρα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Το βρήκατε όλοι παρακαλώ. Στον κατάλογο ψηφοριών. Πολύ ωραία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 2. Και 4. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρινεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5 και 6 από κοινού υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 7 και 8 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 και 10 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία τελική έναρξη ψηφοφορίας 54 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, 0 αποχές. Ωραία λοιπόν. Ολοκληρώθηκε και αυτή η ψηφοφορία και τώρα θα πάμε στην ΕΦΣΑ, στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Τροπολογία 1. Υπέρ αποχές εγκρίνεται. 2 και 3 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 και 5 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφέ Παρακαλώ να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα τη 7 ηλεκτρονικά. Ψήφισατε παρακαλώ όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οκτώ και εννέα μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ηλεκτρονικά παρακαλώ τελική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 50 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, 0 αποχές. Και τώρα συνεχίζουμε με τη Σουηδία. Με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Το βρήκατε? Πολύ ωραία τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 και 3 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 4 και 5 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 και 7 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 50 ψήφοι υπέρ 10 κατά και 1 αποχή και τώρα περνάμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Τραπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 2, ε, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 3 και 4 από κοινού, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 5 και 6 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 και 8 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 9 και η 10 να ελέγξουμε παρακαλώ την 7 και την 8 ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας πέρας απορρίπτεται η 9 και η 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 53 ψήφοι υπέρ, 8 κατά, 0 αποχές. Έτσι χορηγείται και εδώ η απαλλαγή. Και τώρα. So, damit sind wir Και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες μας περνάμε τις πλαστικές σακούλες την έκθεση μακρέτε Άουκεν. Όλοι είσαστε ευπρόσδεξοι για να συμμετέχετε στη συζήτηση. Όσοι δεν, δεν θέλετε να συμμετάσχετε, παρακαλώ γρήγορα και αθόρυβα να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Gut, Wir können starten mit Tagesordnungspunkt 1. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το 21 της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν επιθυμίας της εισηγήτριας να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίθετα με τις συνήθειες μας. Ο κύριος Λάγκεντορφ είναι εδώ και θα πάρει το λόγο. Thank you, uh, Chair. I'll be uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, είναι απλή η πρόταση, ε, δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εισαγωγή, ανταποκρίνεται στις ανησυχίες για την υπερβολική κατανάλωση πλαστικών ουσιών, σακούλες ιδιαίτερα, ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις από πλευράς κρατών μελών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις σακούλες μεταφοράς. Έγινε διαβούλευση, υπάρχει στήριξη για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Αυτό είναι συμβατό γενικά και με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πλαστικά γενικότερα έχει υπάρξει μια μελέτη επιπτώσεων η οποία χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα δεδομένα αν και υπάρχουν και πάρα πολλά κενά βέβαια για τον ακριβέστερο υπολογισμό των αυτών των προϊόντων, τις σακούλες μεταφοράς εννοώ που κυκλοφορούν στην αγορά. Υπάρχουν και αρκετά μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη βέβαια σε σχέση με τα επίπεδα κατανάλωσης. Υπάρχουν χώρες με πολύ χαμηλά επίπεδα, με πολύ ελαφρές σακούλες και μικρού βάρους δηλαδή και υπάρχουν και άλλες με πολύ υψηλότερη κατανάλωση. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να βάλουμε κάποιους στόχους ε, για τη μείωση της χρήσης αυτών των προϊόντων χαμηλού βάρους, αλλά να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να πάρουν κάποια μέτρα μέσω ε, των οποίων να αναφέρουν μετά στην Επιτροπή για να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις. Πιθανώς δηλαδή να επανέλθουμε με άλλες προτάσεις έτσι ώστε να καταλήξουμε κάπου. Η ίδια η πρόταση λοιπόν τροπολογεί την οδηγία για την συσκευασίες, ιδιαίτερα τα άρθρα 2 και 3, όπου περιλαμβάνονται και ορισμοί για τις σακούλες μεταφοράς, τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Τροπολογεί επίσης και συμπληρώνει και το άρθρο 2 για τις συσκευασίες απαιτώντας από τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα μείωσης της χρήσης αυτών των ε, προϊόντων χαμηλού βάρους, πλαστικές σακούλες χαμηλού βάρους, να χρησιμοποιήσουν είτε οικονομικά μέσα είτε μέσα περιορισμού στις αγορές, στις συναλλαγές και να αναφερθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα των άνω μέτρων. Δεν έχω κάτι άλλο, νομίζω είναι απλή η πρόταση, αν και θέτει βέβαια ε, αρκετά προβλήματα. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να ειδωθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μείωσης της νομοθεσίας ε, για τα απόβλητα. Είμαστε σε φάση επανεξέτασης των ισχυουσών ρυθμίσεων για την ανακύκλωση και ανάκτηση. Ξέρετε ο, ίσως ότι αντιμετωπίζουμε γενικότερα το θέμα των πλαστικών αποβλήτων και θα ελέγξουμε εκ των υστέρων τα αποτελέσματα της εφαρμογής των διαφόρων οδηγιών που καλύπτουν τα απόβλητα κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε καλύτερα συμπεράσματα. Η πρόταση αυτή περιορίζεται βέβαια όπως είπα μόνο στις α, α, πλαστικές σακούλες ελαφρού βάρους μικρού βάρους και όπως είπα υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια η στόχη, η αναθεώρηση των στόχων κτλ και επίσης και του θέματος του ευρύτερου της συσκευασίας. Ευχαριστώ κύριε Όλαντορφ. Αυτό. Τώρα φτάνουμε στην κυρία Άουκεν. Έχει το λόγο η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία πράγματι έκανε επιτέλους αυτή την πρόταση είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι ε, έπρεπε να συζητηθεί, είναι μια βασική προτεραιότητα. Εδώ και χρόνια λέγω ότι πρέπει να δράσουμε στον συγκεκριμένο τομέα. Όπως είπε και ο κύριος Λάγκεντορφ υπάρχει μια ευρωπαϊκή μελέτη η οποία υποστηρίχθηκε και από μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία ε, απαιτεί πλέον να αναλυφθεί δράση. Ο κύριος Λάγκεντορφ είπε πως τώρα πλέον έχουμε σαν στόχο ε, τη μείωση των νομικών ρυθμίσεων, ε, του αριθμού των νομικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των αποβλήτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε το περιεχόμενό τους. Απλά η οδηγία για τα απόβλητα δεν είναι επαρκώς φιλόδοξη. Και αυτό το οποίο εκπλήσει είναι ότι στα πλαίσια της ανάλυσης την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθούνται μερικές φορές διαφορετικές κατευθύνσεις. Δηλαδή, λέγεται ότι δεν θα πρέπει να βασιστούμε αποκλειστικά σε αυτήν την αντίληψη η οποία είναι υποτίθεται ιδιαίτερος λεπτομερής και ιδιαίτερος τεχνικοεπιστημονική. Εμείς στην δική μας πάντως πρόταση επιλέξαμε να στηριχθούμε στην ανάλυση, στη μελέτη των επιπτώσεων. Το κάνουμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι οι πλαστικές σακούλες είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ε, στην Ήπειρό μας, ιδιαίτερα στον τομέα της μόλυνσης. Είναι ένα πρόβλημα βέβαια το οποίο επαναλαμβάνω είναι ορατό. Υπάρχουν χωράφια διάσπαρτα με πλαστικές σακούλες σε πολλές περιοχές αυτό είναι κάτι το οποίο θίγει το περιβάλλον και όχι μόνο το περιβάλλον των ε, υπηρετικών περιοχών αλλά και των θαλασσών. Ακόμα και σε χώρες όπως τη δική μου έχουμε μειώσει με την κατανάλωση και την χρήση των πλαστικών αυτών. παρόλα αυτά το πρόβλημα με τις σακούλες παραμένει. Εάν δεν κάνουμε τίποτα είναι σαφές ότι το 2020 θα έχουμε φτάσει τα 110 δις πλαστικές σακούλες το 2020. Νομίζω ότι αυτός ο αριθμός απαιτεί πλέον να το συζητήσουμε. Τι συμβαίνει τώρα με αυτές τις σακούλες. Ξέρετε ότι οι μισές από αυτές τις σακούλες καταλήγουν στις χωματερές. Τις παίρνει ο αέρας, το 40% ε, καίγονται και μόνο το 20% ανακυκλώνονται. Υπάρχει δηλαδή μια σημαντική απώλεια πόρων. Στην έκθεση την οποία σας παρουσιάζω σήμερα και όπως σας προείπα, εγώ ακολουθώ απλά την ανάλυση των επιπτώσεων στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν τρεις βασικές προτάσεις Πρώτον, θα πρέπει να καθοριστούν στόχοι μείωσης. Εμείς θα θέλαμε οι στόχοι αυτοί να είναι πιο ξεκάθαροι. Όταν μιλάμε για μία μείωση κατά 80% της μέσης κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας σε σχέση με το 2010. Αυτή είναι η βασική μας πρόταση. Υπάρχει επίσης και μια άλλη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να καθορίσει μια τιμή πώληση για τις πλαστικές τσάντες σακούλες. Και ταυτόχρονα εμείς προτείνουμε ένα σχετικά αυστηρό αλλά ρεαλιστικό διετές χρονοδιάγραμμα. Να δούμε τι γίνεται βέβαια στα κράτη-μέλη από τη μία μέρα στην άλλη όταν ορίζεται μια υποχρεωτική τιμή πώληση, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν γιατί οι πολίτες, οι καταναλωτές θα βρουν κάποιες άλλες λύσεις για τη μεταφορά των προϊόντων. Πέραν λοιπόν του ότι εμείς ακολουθούμε τις γενικές κατευθύνσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνουμε επίσης και μια σταδιακή κατάργηση της χρήσης της πλαστικής σακούλας. Υπάρχουν ε, μικρά ε, τμήματα των, ε, του πλαστικού που αποτελεί τις σακούλες, τα οποία δεν είναι βιοαναλώσιμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν επιβάρυνση του περιβάλλοντος και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ουσίες οι οποίες λειτουργούν με πολύ αρνητικό τρόπο για την υγεία. Ενθυμίστε την έκθεση πρώτη. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία κινδύνου θα έλεγα εδώ. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σομαρά και να καταργήσουμε επιτέλους τις πλαστικές σακούλες. Στον τομέα των βιοδιασπόμενων υλικών, για να χαρακτηρίσουμε βιοδιασπόμενο ένα υλικό, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια θα πρέπει αυτά τα απόβλητα να μπορούν να εξαφανιστούν εντελώς να απορροφηθούν μέσα σε μια χρονική περίοδο ενός έτους. Οι κανόνες λοιπόν για τον χαρακτηρισμό ενός τέτοιου προϊόντος ως βιοδιασπόμενου πρέπει να είναι ουσιαστικοί κανόνες. Εάν ένα πλαστικό είναι βιοδιασπόμενο και αν πράγματι οι χώρες έχουν νομοθετικές ρυθμίσεις ξεχωρισμένες ξεχωριστές για τα βιολογικά βιοδιασπόμενα πλαστικά προϊόντα, τότε θα μπορούσαμε ίσως ε, τις σακούλες αυτές να τις χορηγούμε και δωρεάν. Να υπάρχει δηλαδή μια απόκληση από την κεντρική ρύθμιση και να χρησιμοποιούνται για ε, προϊόντα υγρά όπως σαν παράδειγμα το κρέας και τα ψάρια αλλά για τα στεγνά προϊόντα όπως τα λαχανικά και τα λοιπά ε, θα πρέπει πράγματι να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να μειώσουν αμέσως την κατανάλωση των πλαστικών. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, χάρτινες σακούλες, ανακυκλώσιμες σακούλες, επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες κτλ. κτλ. Χαίρομαι λοιπόν που θα ακούσω τώρα και τις παρεμβάσεις των υπολείπων εισηγητών, συνεισηγητών και συναδέλφων και ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου. Ελπίζω ότι θα καταθέσουμε τελικές προτάσεις στους εκλογείς μας επαρκής και θα τους αποδείξουμε ότι είμαστε χρήσιμοι. Σας ευχαριστώ κυρία Άουκαν και τώρα να ακούσουμε τους κοιότητες εισηγητές. Καταρχάς, ε, κυρία Μακουνάιτε, έχει το λόγο. Ε, ε, Όταν είδαμε ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε την οδηγία για τις πλαστικές σακούλες, αναρωτηθήκαμε ποιες, για ποιες πλαστικές σακούλες μιλάμε ακριβώς έγιναν πολλές συζητήσεις. Μιλήσαμε για τις σακούλες μίας ή πολλαπλών χρήσεων για να δούμε αν Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ε, ελαφριές ε, σακούλες που χρησιμοποιούμε για ξηρά προϊόντα και λαχανικά ή αν έχουμε κατά νου τις ε, σακούλες που χρησιμοποιούμε όταν βγαίνουμε από τα καταστήματα τα καταστήματα για τα παπούτσια, τα ρούχα. Είναι ευρύτατο το φάσμα ε, των ε, ε, ειδών που, πλαστικής σακούλας που υπάρχουν. εάν μπω στη θέση του καταναλωτή θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια και πραγματικά ελπίζω ότι θα είναι αποτελεσματική συνεργασία μας. Θα πρέπει να έχουμε διάφορες κατηγορίες 10, ε, 50 μάικρον ε, για, όπως σας είπα, για νοπά προϊόντα, ξηρά ή υγρά ε, και ξαναλέω πως το βασικότερο πρόβλημα είναι οι μικρότερες σακούλες σε 10 μάικρον, διότι εγώ προσωπικά τις μεγάλες σακούλες τις χρησιμοποιώ πολλές φορές και όχι μόνο μία. Είναι πιο μακρύβιες, ας το πω έτσι. Ενώ οι ελαφριές ε, μικρές σακούλες ε, δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα και το αναφέρει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρότι μας λέει ότι δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Τι συμβαίνει λοιπόν για την ανακύκλωση. Έχουμε διάφορα προβλήματα. Πρώτο ε, πρόβλημα ο τρόπος συλλογής. Υπάρχουν λοιπόν εναλλακτικέ λύσεις. Μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο χρήση ε, χάρτινων σακουλών ε, και όπως ε, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία στη διάθεσή μας τόσο ώστε να κάνουμε μια σωστή επιλογή και να προτείνουμε τις εναλλακτικέ λύσεις. ή για να καταλήξουμε σε αυτή την κατάταξη. Αν θα έχουμε κατηγορίες με μικρές και μεγάλες σακούλες ή θα έχουμε μία ενιαία ε, ομάδα. Επίσης, υπάρχουν διαφορές ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, όχι μόνο ως προς την νομοθεσία για τις ακουλές, αλλά και ως προς τις περιβαλλοντικές ε, ανησυχίες. Οι ελαφριές ακούλες παράγονται κυρίως στην Ασία και ε, εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο συμβαίνει με τις μεγαλύτερες ακούλες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τον τόπο προέλευσης Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ε, απαγόρευσης ε, κάποιων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, για την κατασκευή ε, της σακούλας. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για τη συλλογή επίσης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη και την ανακύκλωση. Και ποιο θα είναι το σημείο εκείνης το 2010, όπως αναφέρεται δεν θα συμφωνήσω, ε, μιλώντας φυσικά για τον υπολογισμό ε, των ποσοστών χρήσης ε, στα κράτη-μέλη. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί μια εντατική εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού και των καταναλωτών για τη χρήση ούτως ώστε να καταλάβουν πόσο επιβλαβείς είναι οι πλαστικές σακούλες για το περιβάλλον. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, ε, μαρακινηθούν οι καταναλωτές ε, ε, να χρησιμοποιούν περισσότερες φορές τις σακούλες. Τώρα επιστρέφοντας σε αυτά τα ποσοστά μείωσης της χρήσης, δεν μπορούμε να, φυσικά να επιδιώξουμε απαγόρευση αυτού του προϊόντος γιατί γιατί το χρειαζόμαστε για λόγους συσκευασία. Ε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε μέσα σε λίγα χρόνια να επιτύχουμε τόσο υψηλά ποσοστά μείωση όπως το 80%. Ε, ίσως όμως αυτό το 80% υπολογίστηκε με γνώμονα το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ε, με βάση τα εθνικά ποσοστά. Πιστεύω πως ε, θα κατατεθούν πάρα πολλές τροπολογίες, θα γίνουν ευρύτερες ε, συζητήσεις. Παρότι η Επιτροπή μας λέει ότι είναι απλό το κείμενο, δεν θα συμφωνήσω, παρόλα αυτά πιστεύω και ελπίζω ότι θα βρούμε ε, ικανοποιητικές λύσεις. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτές οι σακούλες σχεδόν παντού είναι δωρεάν. Και στην Ολλανδία πάντα σε ρωτάνε αν θέλεις ε, τη σακούλα. Ε, και φυσικά όλοι απαντάνε ναι. Είναι απλό. Το 2010 189 τέτοιες σακούλες ε, χρησιμοποίησε. Κοιτάξτε πόσες μέρες έχει ο χρόνος Κάθε δηλαδή δύο ημέρες ουσιαστικά έχει κανείς μια νέα σακούλα πλαστική που χρησιμοποιεί. Και βλέπουμε ότι οι πολιτικοί στον τομέα αυτό μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί είναι δωρεάν αυτή τη στιγμή οι σακούλες και όπως μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν αναφέρεται, δεν ε, συμπεριλαμβάνεται το εξωτερικό κόστος, ε, η πρώτη ύλη, η μόλυνση των, του περιβάλλοντος σε μακρινά νησιά. Ξέρουμε όλες τις φωτογραφίες με τους ε, γλάρους που είναι πνιγμένοι στο πλαστικό. Και βλέπουμε ότι αυτές οι πολιτικές μπορούν να λειτουργήσουν και μιλάμε για πολλά τέτοια θέματα που άπτονται των καταναλωτών και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Υπάρχουν χώρες που έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα, η Φιλανδία, η Δανία, όπου χρησιμοποιούνται και 500 φορές λιγότερα, λιγότερες πλαστικές σακούλες. Χώρες δηλαδή που δεν ε, αποδεχόμαστε μία σακούλα κάθε δύο μέρες, αλλά μία φορά, για παράδειγμα, την εβδομάδα. Το σημαντικό είναι ότι ο πολίτης το δέχεται αυτό, γιατί είναι και πολύ άνετο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στρέφεται κυρίως στις ελαφριές ε, πλαστικές σακούλες για να περιορίσει τον αριθμό των σακούλων αυτών που καταλήγουν στους ωκεανούς. Και για παράδειγμα στην ταινία American Beauty βλέπουμε επί 10 λεπτά μια σακούλα πλαστική που ανεμίζει και περιφέρεται. Πάντα λοιπόν είναι ένα θέμα αυτό και αν ε, καταφέρναμε να τις κάνουμε διαλυτές αυτές τις σακούλες, ε, θα είχαμε ανακαλύψει το από του Κολόμβου. Αλλά δεν θα διαλύονταν τελικά και στη θάλασσα. Και αυτές οι βοαποδομήσιμες είναι καινούργιο μοντέλο. Ίσως εκείνα είναι το μέλλον, αλλά στην παρούσα φάση έχουμε χαθεί σε ένα δάσος από ορισμούς βιοαποδομήσιμων που τελικά δεν είναι βιοαποδομές, είναι βιό ε, ε, διασπόμενες, ένα σωρό ορισμούς έχουμε και θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Πρόντι που μας παρέχει διάφορους αποδεκτούς ορισμούς ό,τι αφορά την κομποστοποίηση. Να σκεφτούμε και την καινοτομία και την επένδυση σε μελλοντικέ σακούλες, σακούλες που είναι βιοδιασπόμενες και στη θάλασσα υποφυσικές συνθήκες, γιατί συχνά, μάλλον κυρίως ε, μιλάμε σε όλο αυτό το δάσος και στο χαμό των ορισμών, μιλάμε πάντα για βιομηχανικά διασπόμενες, για βιομηχανικά σακούλες σε οι 20 εβδομάδες θα πρέπει να διασπώνται και να επιστρέφονται και να επανέρχονται τα συστατικά του στο περιβάλλον. Δεν είμαι ιδιαίτερα ενθουσιώδης για ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογή. Έχουμε ένα σύστημα συλλογή και δεν θέλουμε να γίνει ο κάθε πολίτης εμπειρογνώμονα σε θέματα πλαστικής σακούλας. Καλά θα ήταν, αλλά δεν γίνεται. Ενδεχομένως φορολόγηση στα ταμεία να επιβάλλεται ένα τέλος σε ό,τι αφορά τις πιο ε, χοντρές σακούλες, τον οποίων το πλεονέκτημα είναι ότι δεν ε, ε, ανεμίζουν τόσο εύκολα, δεν φεύγουν και χάνονται και καταλήγουν στη θάλασσα τόσο εύκολα. Και νομίζω ότι μία τέτοια σακούλα θα πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον 125 φορές, θα πρέπει να είναι ανθεκτική. Να πω ότι δεν είμαι υπέρ της εξέρεξης για τις μικρές τέτοιες σακούλες, η συγγήτρια λέει ότι είναι απαραίτητες για τη συσκευασία διαφόρων τροφίμων. Αλλά κοιτάξτε, αυτές είναι οι πιο επιζήμιες σακούλιτσες. Να δούμε λοιπόν πως υπάρχει κάποια άλλη λύση από το να εξαιρεθούν. Τέλος, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι σημαντικά. Να σας πω το εξής. Αν, αν πούμε ότι οι βοηδιασπόμενος είναι το μέλλον, ο πολίτης δεν θα να γνωρίζει απαραίτητα γιατί τελικά αν ο πολίτης προσπαθήσει να κάνει κομποστοποίηση μια σακούλας που δεν ενδείκνεται, τελικά θα έχει πρόβλημα, θα έχουμε παραπάνω προβλήματα. Ίσως λοιπόν να σκεφτούμε και ένα σύστημα επισήμανσης της σακούλας. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και είμαι βέβαιη ότι έτσι θα πετύχουμε μείωση της πλαστικής σακούλας και της χρήσης της στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μερκής ο κύριος Μπραντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την συνεισφορά του. Θα πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερο ευτυχής που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε το θέμα της πλαστικής σακούλας και δεν περίμενε όλες τις συνολικές προτάσεις για τα απόβλητα. Καθυστερήσαμε όμως αρκετά χρόνια, είμαστε κοντά στις εκλογές και δεν θα μπορέσουμε εμείς να κλείσουμε το θέμα πριν από τις εκλογές. Θα μπορούσε να έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και δύο χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία μπορούμε εύκολα ε, να λύσουμε. Είναι ένα φρούτο που κρέμεται χαμηλά στο δέντρο. Στο βορρά της Ευρώπης το 70% των πλαστικών αποβλήτων προέρχεται από τις σακούλες. Πρέπει λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα όπως δείχνουν περιπτώσεις όπως η Δανία, η Ιρλανδία και ακόμα και κάποιες κινέζικες επαρχίες. Δεν είμαστε δηλαδή και πάρα πολύ προχωρημένοι θα έλεγα σε σχέση με άλλες χώρες. Έχουμε πλέον μία πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν υπάρχει ένας δεδομένος τελικός στόχος. Από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δείχνει να θέλει να ενοχλήσει και ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να πιέσουν ε, στον τομέα ε, τον οικονομικό αλλά και τον περιβαλλοντικό. Το είδαμε αυτό σήμερα και για το πακέτο το κλιματολογικό. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση του εισηγητή μας, της εισηγητριάς μας μάλλον, της κυρίας Άουκεν, η οποία θέτει το στόχο του 80%. Πρέπει να είμαστε τόσο φιλόδοξοι όσο προτείνει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο τελικά να πετύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο. Λοιπόν, ένα από τα βασικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα των ορισμών της πλαστικής σακούλας. Απαιτείται εδώ περισσότερη λεπτομέρεια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προτάσεις AUKEN. Τα 10 μικρών τα οποία αναφέρει η κυρία Άουκεν σαν μέγιστο ε, βάρος νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι οι σακούλες τις οποίες παίρνει κανείς τον χασάπι σαν παράδειγμα θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις προτάσεις της. Εγώ δεν ελπίζω να προτείνει την εξαίρεση της σακούλας την οποία παίρνει κανείς στην αγορά για να βάλει τα λαχανικά του και τα υπόλοιπα αφρούτα του. Δεν θα ήθελα εδώ να υπάρξουν εξαιρέσεις για τα λαχανικά παρά μόνο για το κρέας. Λοιπόν αυτά τα 10 μικρών. Το όριο είναι κάτι το οποίο θεωρείται σωστό και είναι εφικτό γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, για το οποίο θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των καρκι... Το θέμα των καρκινογόνων ουσιών είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στα υπόλοιπα τμήματα της ε, ισχύουσας αλλά και προτινόμενης νομοθεσίας. Θέλω να επιταχύνουμε τη διαδικασία εδώ και θα ήθελα να αποφύγουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και να καταλήξουμε στις διαπραγματεύσεις αυτές ε, με ε, πάρα πολύ μεγάλη απώλεια χρόνου σε τέτοιου είδους θέματα. Πάντως επαναλαμβάνω ότι αν ε, γλιτώσουμε το 70% των πλαστικών που καταλήγουν στις θάλασσές μας, τότε πράγματι θα έχουμε κάνει το πάρα πολύ, κάτι το πάρα πολύ θετικό και θα προχωρήσουμε γρήγορα. Er Ευχαριστώ λέει κυρία Όκεν, θα μιλήσω σουηδικά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να... Η κυρία Ρόσμπαχ, συγγνώμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους ε, που σχολίασαν όλα αυτά τα επιμέρους σημεία. Θα διαφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας λέει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και καθόλου περίπλοκο αυτό το ζήτημα. Θα διαφωνήσω κάθετα. Χαίρομαι επιτέλους που έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, τουλάχιστον επιτάπητος, ούτως ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα πρωτού εκπνεύσει η προθεσμία που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα συμφωνήσω επίσης με τους συναδέλφους ε, που μας είπαν ότι λυπούνται διότι ε, καθυστέρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πάρα πολύ με την πρόταση. Ναι, θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε την κατάργηση της σακούλας. Μα δεν είναι ρεαλιστικό, δεν μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό από τους καταναλωτές. Εάν επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο, ε, θα έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν περισσότερο άλλα ε, μέσα συσκευασία. Δεν είναι εύκολο να ξεφορτωθούμε ε, την πλαστική σακούλα. Υπάρχουν και άλλα μέσα συσκευασία από πλαστικό ή από χαρτί ή από πεπιεσμένο χαρτί. Υπάρχουν διάφορα μέσα Και μην ξεχνάμε ότι ακόμη και το χαρτί δημιουργεί περιβαλλοντικό πρόβλημα. Πέραν αυτού χρησιμοποιούνται και πολλές χημικέ ουσίε για την παραγωγή χαρτοπολιτού. και γνωρίζετε πως ε, στην βιομηχανία χάρτου χρησιμοποιούνται ε, πολλοί άριθμες ε, χημικές ουσίες. Λοιπόν, δεν είναι μία μόνο η λύση. Θα πρέπει να διερευνήσουμε όλες τι εναλλακτικέ οδού που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Έχω ήδη λάβει διάφορα ε, αιτήματα, αλλά και ε, με έχουν πλησιάσει πάρα πολύ κρούντας τον κόδωνα του κινδύνου, ε, φυστώντας την προσοχή μου σε διάφορα κρυμμένα προβλήματα. Είναι πολυδιάστατο το ζήτημα. Το βιοδιασπόμενο πλαστικό είναι ένα άλλο σημείο που ε, σχολιάστηκε στη συζήτηση. Δεν μπορούμε ε, να ε, επιλέξουμε ε, την ε, χρήση και μόνο αυτού του βιδιασπόμενου πλαστικού, διότι για την παραγωγή του πάλι χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες. Δεν είναι πανάκια λοιπόν, ε, βιοδιασπάται ναι μεν, αλλά σε μικρά μόρια τα οποία απορροφούνται από το περιβάλλον, δεν εξανεμίζεται, δεν ε, εξαφανίζεται αυτό το πλαστικό, μετατρέπεται απλώς σε πολύ μικρά μόρια. Ε, άλλο πρόβλημα είναι τα απόβλητα. Διαφέρουν πολύ τα εθνικά συστήματα συλλογής και διάθεσης αποβλήτων. Στη δική μου χώρα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά ξέρω ότι σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν καν συστήματα συλλογής για τις ακούλες Θα πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε και μία εναρμόνιση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσπαθήσουμε, διότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια στον τομέα αυτό, δεν έχουν αναλάβει κανένα μέτρο. Και γι' αυτό σας λέω πρέπει να είναι πολλαπλή η στόχη μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή λύση. Ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η μέγιστη δυνατή προσπάθεια που μπορεί να κάνει ένα κράτος μέλος. Άλλη κατάσταση στη Δανία, άλλη στη Γερμανία, άλλη σε άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε οι χώρες που δεν έχουν κάνει προς το παρόν πολλά πράγματα να δράσουν επιτέλους. Ας μην τιμωρήσουμε όμως τις χώρες που έχουν ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Στη χώρα μου, ξαναλέω, εδώ και καιρό ε, συνειδητοποιήσαμε ότι αν ζητήσει κανείς 50 λεπτά ε, του ευρώ στο καταναλωτή για να πάρει τη σακούλα, θα βρει εκείνος άλλο τρόπο για να μεταφέρει τα ψώνια στο σπίτι του για να μην καταβάλει το αντίτιμο. Ε, δεν έχουμε πλαστικές σακούλες, ε, ε οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ε, χαρτόκουτα ή τσάντες ε, που χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν τα ψώνια και να τα ξεφορτώσουν ε, στο παγκάζ του αυτοκινήτου τους στη συνέχεια. Δεν είναι ε, καλό να απορρίπτονται οι πλαστικές σακούλες στο περιβάλλον. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε στους καταναλωτές. Ε, το πλαστικό πρέπει να το ξαναχρησιμοποιούμε, δεν είναι απόβλητο. Θα πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουν οι καταναλωτές ε, και να καταλάβουν ότι πρέπει να επιδιώκουν το μέγιστο αριθμό χρήσεων κάθε πλαστικής σακούλας διότι είναι ε, ένας πόρος, δεν είναι ένα απόβλητο. Λοιπόν, θα πρέπει να διαθέσουμε και τα να κονδύλια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών θα χρειαστούμε την πιο ρεαλιστική και την πιο ευέλικτη δυνατή λύση. Προσβλέπω στην ε, συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα περάσουμε στους επόμενους ομιλητές, ε, λοιπόν. Δύο λεπτά έκαστος, ε, παρακαλώ. Μην υπερβείτε το χρόνο σας και κοιτάζω καλά-καλά την Κρίστα Κλάς, πρώτη και καλύτερη. denke man muss schon auch differenziert sehen und ich Ευχαριστώ είναι απλά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει, υπάρχουν πολύ διαφορετικές χρειές σε όλες αυτές τις επιμέρους ιδέες. Νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τους καταναλωτές. Ε, υπάρχουν ε, κάποια μέσα συσκευασία που είναι απαραίτητα για κάποια προϊόντα και φυσικά ε, δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ευθύνη των καταναλωτών, είναι και θέμα κόστους. Ε, στα, για τις πλαστικές σακούλες σε ε, κάποια κράτη-μέλη υπάρχει ένα αντίτιμο για τις πλαστικές σακούλες και εκεί ε, μειώνεται η χρήση. Και η μείωση κατά 80% ουσιαστικά είναι απαγόρευση. Δεν μπορώ λοιπόν να συμφωνήσω με αυτό. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις σακούλες. Άλλοι τις δίνουν δωρεάν, δεν τις χωρίζουν. Άλλοι ζητούν να πληρώνονται και να ε, απορρίπτονται με ξεχωριστό τρόπο και στη Γερμανία για παράδειγμα υπάρχει ένα σύστημα ε, όπου χωρίζονται και απορρίπτονται ξεχωριστά οι σακούλες και έτσι δεν επιβαρύνεται ο καταναλωτής με την απορρίψή τους. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε και να προωθήσουμε αυτά τα συστήματα και αυτούς τους μηχανισμούς. Υπάρχουν και καινοτόμες ε, τέτοιες μέθοδοι και μπορεί έτσι να δημιουργηθούν και θέσεις εργασία στην Ευρώπη. Ε, επαναχρησιμοποίηση, μείωση της χρήσης και πολλαπλές χρήσεις, βιολογική διασπασιμότητα, βιολογική ε, βάση bio-based, biodegradable. Νομίζω ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν αυτά. Και επίσης, όταν μιλάμε για πλασικό, νομίζω ότι παραπλανούμε τον καταναλωτή όταν μιλάμε για βιολογική οτιδήποτε διάσπαση, βάση. Γιατί η διαδικασία αυτή εξακολουθεί να παίρνει πάρα πολύ καιρό και αυτό δεν μπορεί από οικολογικής άποψης να βγάζει νόημα. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν μια αποφασιστική προσέγγιση. Θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υποβάλουμε σχετικές προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι το πλαίσιο το οποίο συζητάμε αναφέρεται στα λεγόμενα παραδοσιακά πλαστικά διότι είναι αυτά που έχουν ε, την μεγάλη σταθερότητα, διάρκεια δηλαδή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο περιβάλλον. Θα ήθελα όμως εδώ να θυμίσω ότι ειδικά στην Ευρώπη έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος για την παραγωγή πλαστικών ουσιών οι οποίες να είναι ουσιαστικά βιοδιασπόμενες και να μπορούν να γίνουν και να συμπεριληφθούν σε κομπόστ. Περιλαμβάνουν λοιπόν το πλεονέκτημα να χρησιμοποιούνται χωρίς να υπάρχουν οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για το περιβάλλον. Θα ήθελα λοιπόν να μπορέσουμε να προβούμε στην συγκεκριμένη ε, διάκριση. Γιατί μιλάμε για πλαστικές ουσίες, οι οποίες έχουν ε, βιολογική βάση, έχουν δημιουργηθεί δηλαδή από φυτικά κυρίως υλικά. Θεωρώ λοιπόν ότι τα λεγόμενα bio-based που βασίζονται δηλαδή σε βιολογικά υλικά δεν σημαίνει ότι είναι και βιοδιασπόμενα. Όμως οι τσάντες αυτές, οι σακούλες αυτές μπορούν να είναι βιοδιασπόμενες, μπορούν να γίνουν κοπόστ, και μπορούν επίσης, μπορούμε συνεπώς να βελτιώσουμε εμείς την μεταφορά των υγρών ή φρέσκων προϊόντων που απαιτούν πλαστικές σακούλες για τη μεταφορά τους. Μπορούν να καλύψουν λοιπόν τις ανάγκες αυτές οι συγκεκριμένες σακούλες. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες βιοδιασπομένων πλαστικών που θα πρέπει να αποφύγουμε γιατί δεν είναι ουσιαστικά βιοδιασπόμενες αλλά διασπώνται σε μικρότερα τμήματα και μόρια τα οποία τελικά μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι πιο επικίνδυνα. Έχουμε λοιπόν τα επίπεδα τα απαραίτητα, έχουμε τις βιομηχανικές μονάδες έτσι ώστε οι σακούλες αυτές οι οποίες ε, έχουν μια κάποια θετική θα έλεγα πλευρά στην καθημερινότητά μας ε, πρέπει να μπορούν οι πολίτες να τις χρησιμοποιούν γιατί δεν έχουν συνέπειες σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Ο Καλ Χάιντς για δύο λεπτά. Ναι, πολλά ακούσαμε και δεν θα ήθελα να επαναληφθώ και πολλά είναι σωστά. Η κυρία Άουκεν ε, πρέπει να πω ότι έχει υποβάλει ένα καλό έγγραφο. Το 80% είναι σκληρό στόχος. Εμείς φοβόμαστε, φοβάμαι λίγο όταν ξεκινάμε από τους καταναλωτές. Γιατί, αγαπητή Επιτροπή, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για κάποια πράγματα επί της πολιτικής, με κάποια ιεραρχία, με πολλές ε, εναλλακτικές λύσεις γιατί δεν έχουμε ε, ε, οδηγία για τους χιτά. Το βλέπουμε αυτό και στη Γερμανία και στη Δανία και σίγουρα και σε άλλες χώρες. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν είμαστε τέλειοι, όχι βέβαια. Αναρωτιέμαι όμως, αυτοί που ζητούν τις ε, σακούλες στον χασάπι, αλλά όχι στην αγορά, στη λαϊκή. Ε, μα πώς να το ξεχωρίσει αυτό ο νομοθέτης. Νομίζω ότι χρειάζεται ε, μία αντικειμενική πολιτική για την ανακύκλωση. Είμαστε ούτε καν στη Γερμανία. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στη συλλογή, αλλά όλα τα βάζουμε σε έναν, ε, σε, ε, έναν καυστήρα όλα αυτά μαζί. Αυτό λοιπόν ε, είναι το πρόβλημά μου. Κατά τα άλλα συμφωνώ με την έκθεση και με ικανοποιεί αγαπητέ στην Πρόντι. Αυτό το βιοπλαστικό έχει τόσες πολλές διαφορετικές πτυχές. Δεν ε, βιοδιασποώνται, κομποστοποιούνται αυτές, ε, αυτά το πλαστικό. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και δεν είναι λοιπόν αυτό η απάντηση Χρειάζεται λοιπόν πολύ πιο ακριβής πολιτική για, τις, ε, ε, για τους χώρους απόρριψης προκειμένου να μην καταλήξουμε σε μια κλασική πολιτική καύσης. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι προσωρινό. Χρειαζόμαστε μια νέα ιστορική πολιτική εξέλιξη στον τομέα αυτό και όχι μια πολιτική απαγόρευση απλά. Σας ευχαριστώ. Αντιγέσκου και Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Plastic subțiri și doresc să-i mulțumesc și eu, doamnei raportor, pentru munca depusă. Am avut ocazia... Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι πλαστικές σακούλες είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή Intriga pe cetățenii europeni și cred că Απαιτείται να υπάρχει μεγαλύτερη, καλύτερο αν θέλετε νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την κατανάλωση των πλαστικών αυτών. και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουν τους στόχους τους για τις πλαστικές σακούλες. Θα πρέπει να λύσουμε λοιπόν επιτέλους το θέμα αυτό της ε, ε, άπαξ χρήσεως των πλαστικών για μεταφορά προϊόντων. Οι κοινοτικές αρχές όπως επίσης και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες οι οποίες ε, υπάρχουν σήμερα και πράγματι θα πρέπει να αποφύγουμε ε, την, τις τσάντες αυτές που αποτελούνται από πλαστικό το οποίο απλά διασπάται σε πολύ μικρότερα τμήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει κυρία Βέστλοντ, ευχαριστώ επίσης και την εισηγήτρια για την πρότασή της. Είναι μια πρόταση πάρα πολύ φιλόδοξη όταν οι πλαστικές σακούλες εισήχθησαν στην αγορά η επιτυχία τους ήταν τεράστια και αντί να κουβαλάμε ε, τα βάρη μας στον ώμο μας αρχίσαμε να κουβαλάμε φυσικά με τα χέρια μας και αυτό έχει συνέπειες βέβαια πολύ σημαντικές για τη σπονδυλική μας στήλη. Αυτό είναι θέμα πολιτιστικό και νομίζω ότι πρέπει να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο. Στην Κίνα δεν είδα κανέναν να κουβαλάει ε, πλαστικές σακούλες ή να κυκλοφορούν ε, πλαστικές σακούλες ε, γιατί τις ανακυκλώνουν και δεν φαίνονται. Στην Τινησία πάλι είναι μια χώρα η οποία ζει με τις πλαστικές σακούλες. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τους κινδύνους για το περιβάλλον και θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε πώς μπορούμε να πείσουμε τους νέους, να τους δείξουμε στους νέους το τι είναι μοντέρνο, τι είναι cool σε εισαγωγικά. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών ε, κατά 80%. Αυτό όμως είναι δύσκολο γιατί αυτό θα θίξει φυσικά και αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τις σακούλες αυτές και που παράγουν τις σακούλες αυτές απαιτούνται μελέτες, απαιτούνται νέα υλικά, απαιτούνται αξιολογήσεις. Εγώ δεν είδα καμία ουσιαστική έρευνα και αξιολόγηση σχετικά με τις ανάγκες των νέων. Δεν είδα καμία ε, μελέτη και αξιολόγηση των βιομηχανικών συνεπειών ενός τέτοιου μέτρου. Στην Σλοβενία σαν παράδειγμα δεν βρίσκει κανείς εύκολα πλαστικές σακούλες, πρέπει να τις πληρώνει, δεν είναι ποτέ δωρεάν αλλά αυτό δεν αρκεί. Η ενημέρωση και η συνειδητοποίηση στην Σλοβενία γίνονται με σωστό τρόπο. Ευχαριστώ. Sorry. Благодаря, господин председател. Κυρία Λουμπιτσέβα говорим за опасности от употреба на пластмасовите турбички, но трябва да сме много откровени и да си признаем, че до преди няколко години тяхната употреба... Συγγνώμη, αλλά έχουμε ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό, λέει ο πρόεδρος. We have to close the meeting. No. so, can we start again? Πρέπει να ξαναρχίσετε, λέει ο πρόεδρος, την κυρία Λιούπτσεβα. Сега наред ли е? Okay. Колеги, а, днес говорим за ограничаване а, и за опасност. Συνάδελφοι, σήμερα συζητούμε για τους κινδύνους που επισύρει η χρήση της πλαστικής ε, σακούλας ε, με χερούλια. Ε, κάποτε θεωρούσαμε μεγάλο προνόμιο τη χρήση αυτή της σακούλα, διότι μας διευκόλυνε το ότι μας δημιουργεί πρόβλημα αυτή η σακούλα σήμερα, σημαίνει ότι πρέπει ε, ε, να αλλάξουμε το, τις συνήθειές μας και να μειώσουμε την κατανάλωση. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό, ενημερώνοντας τους πολίτες ε, για τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής της πλαστικής σακούλας. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας επίσης. Αυτό είναι κάτι δύσκολο. Ε, χρειάζεται αρρωγή των νέων. Ε, οι νέοι υιοθετούν διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με τους πιο ηλικιωμένους ως προς τη δυνατότητα βιοδιάσπασης της πλαστικής σακούλας οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε αυτή την διάκριση ανάμεσα στις μικρές και μεγαλύτερες ε, πλαστικές σακούλες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και για λόγους ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις. αυτές τα θέματα ανταγωνισμού δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα σε κάποιες χώρες. Υπάρχουν πάντως ελιπέστατες πληροφορίες για τους καταναλωτές σε σχέση με τη βλαστική σακούλα και δεν ξέρουν καν πώς να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα σε μια διασπόμενη και μια μη βιοδιασπόμενη σακούλα. Θέλουμε λοιπόν, όπως έλεγα, να μειώσουμε, να περιορίσουμε τη χρήση ε, πώς αλήθεια μπορούμε να το πετύχουμε αυτό δεδομένων των ε, διαφορών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε μία ενιαία πολιτική η οποία προϋποθέτει πολύπλοκα μέτρα που αφενός θα ρυθμίζουν την κατανάλωση αφετέρου θα φροντίζουν για την ενημέρωση του καταναλωτή. Ξαναλέω, δεν ε, έχουν σωστή ενημέρωση οι καταναλωτές για το πόσο επιζήμιες είναι οι σακούλες, κυρίως δε οι σακούλες των 10 μάικρων για το περιβάλλον. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση πρέπει να συλλέξουμε ακριβέστερα στοιχεία. Ε, ε, ε, αφήστε δε που η συλλογή συνεπάγεται και άλλους κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν το σύνολο αυτών των προβλημάτων να το αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε ποιες είναι οι πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ ο Κάρος Σλούτερ. Ε, ευχαριστώ. Νομίζω α, υπόθηκαν όλα από τους συναδέλφους, ε, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ εγώ στο όριο των 15 μάικρων κάτω αυτού του ορίου θεωρείται κανόνας ότι είναι βιοδιασπόμενη η σακούλα. Τι σημαίνει όμως βιοδιασπόμενος. Ε, ε θεωρούν κάποιοι ότι αν ε, διασπάτε κάτι και οξυδώνεται αλλά αφήνουν ε, 10.000 ε, τμήματα της χιλής μόρια μετά την υποδιάσπαση τότε εκπέμπεται παρόλα αυτά διοξίδιο του άνθρακα. Δεν ξέρω λοιπόν. Ε, κάποιε κάποιες βιοδιασπόμενες σακούλες επίσης περιέχουν και κάποια πλαστικά που δεν είναι βιοδιασπόμενα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε καλό ορισμό τόσο ώστε να είναι πλήρως ε, βιοδιασπόμενες οι σακούλες. Ε, κάτι άλλο τώρα. τι συμβαίνει μετά αν ε, καταλήξει σακούλα στη χωματερή όπου ε, μετατρέπεται σε ένα αναερόβιο περιβάλλον και παράγει μεθάνιο, τότε ε, παράγουμε εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου. Πρέπει να δούμε τι θα τι κάνουμε τις ε, βιοδιασπόμενες. Μπορούμε να ζητήσουμε πάντως για τις λεπτές και ελαφριές ε, ότι πρέπει να είναι πλήρως ε, βιοδιασπόμενες και σίγουρα θα πρέπει να πληρώνουν όλοι για τη χρήση τους γιατί έτσι θα το σκέφτονται καλύτερα πρωτού τους χρησιμοποιήσουν. Πριν από 40 χρόνια ήταν στο λιανεμπόριο, στην Ένωση Λιανεμπόρων ο πατέρας μου και έγινε μια τέτοια απόπειρα. Τότε γίνανε διαδηλώσεις κατά αυτής της καινοτόμου ιδέας. Τώρα όλοι το θεωρούν είναι φυσιολογικό. Εντάξει, θα ακούσουμε τι κριτικέ, θα παραπονεθούν όλοι για κάνα δύο εβδομάδε και μετά θα το θεωρήσουν όλοι φυσιολογικό. Ε, ε υπάρχει, εγώ κάνω επίση μια καμπάνια και για τι ε, υφασμάτινε τις σακούλες. άμα με επικοινωνήσετε μαζί μου, να σας δώσω και μία. Ευχαριστούμε. Ε, Πίτερ ε, Λίζε και νομίζω μετά θα, θα συνεχίσουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε με τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Λίζε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Αόκεν. Εγώ ε, μίλησα με αυτούς τους αρμόδιους φορείς για τη συλλογή των αποβλήτων ε, στην εκλογική μου περιφέρεια. Είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ψηφοφόρους μας. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν θα ταχθώ υπέρ μιας απαγόρευσης. Ακόμη και οι πράσινοι ε, στη Γερμανία δεν θεώρησαν ότι η ιδέα της απαγόρευσης ε, στέφθηκε με επιτυχία. Η κυρία Κλάς ε, είχε την καλύτερη ιδέα, ένα μικρό αντίτιμο για μικρές σακούλες. Είναι αυτό που θα έπρεπε να προτιμήσουμε. Τι γίνεται μετά τη χρήση της σακούλας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό δε, διότι ε, εκεί αρχίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το να έχουμε τώρα ένα νέο στόχο μείωσης 80%, ε, κατά 80% είναι σφαλμένη οδός. Χρειάζεται ε, κατακεφαλή υπολογισμό, διότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, σε κάποιες χώρες, παραδείγματο χαρή, είναι ήδη πολύ περιορισμένη η χρήση. Για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να είναι πιο ρεαλιστική η στόχη. Έχω και ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα η νομική βάση είναι προβληματική διότι χρησιμοποιούμε τη νομική βάση για τις είναι οργανώσεις ε, αγοράς. Τα κράτη-μέλη δηλαδή πρέπει να κάνουν αυτό ε, ή εκείνο, να αναλάβουν κάποιο μέτρο. Όμως πέρα από την απαγόρευση, τι συμβαίνει όταν σε κάποιες χώρες θα έχουμε απαγόρευση 11 παραδείγματο χάρη και σε άλλες θα έχουμε αντίτιμο ε, για την χρήση της σακούλα. δεν θα υπάρξει εναρμόνιση. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω... Είναι, είναι όντω έτσι ότι στην, ε, ισχύει ότι στην Κίνα, για παράδειγμα, υπάρχουν ειδικά τέλη και τι γίνεται και με, τις, ε, με το βιολογικό χαρτί. Ένα τελευταίο επιχείρημα οι λομπίστες υπέρ της πλαστικής σακούλας ε, να μην ανατρέψουν για την πραγματικότητα. Είπαν ότι ε, για τις σακούλες αυτές δεν πρέπει να τις πλένει κανείς ε, για να μην κολλήσει οι ασθένειες και να μην μου χλιάσουμε το καθεξά, να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης. Κοιτάξτε, Υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία είναι σοβαρά σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς ε, των, ε, της σακούλας αυτής, αλλά αυτό το επιχείρημα δεν βρίσκω ότι είναι ε, σοβαρό. Ναι, δηλαδή ότι η ημερομηνία ανάλωσης είναι πέντε ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Ε, η κυρία Σοφία Οκονή και μετά τον Αρσένης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούστηκαν πολλά πράγματα και γι' αυτό θα ήθελα τρία μικρά στοιχεία να καταθέσω. Το πρώτο, να πω ότι όπως είπε και ο Φλόρεντς, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ορισμένες εθνικές ρυθμίσεις οι οποίες ε, μειώνουν ε, με σημαντικό ποσοστό την κατανάλωση των ε, ε, των, αυτών των πλαστικών μέσω ε, και της δημιουργίας ε, προϊόντων με βιοδιασπόμενα υλικά. Πρέπει να δούμε εδώ τι γίνεται με την καινοτομία και την έρευνα. Εγώ πήγα και επισκέφτηκα τον σταθμό καθαρισμού υδάτων των Βρυξελών που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη Εκεί ανέλησαν τα ύδατα που εξετάζουν και είδαν ότι υπήρχαν ε, πολυμερισμένα τμήματα που συνδέονται με τις πλαστικές σακούλες. Βρήκανε ένα βακτηρίδιο το οποίο ε, απορροφά αυτού του είδους ε, τα προϊόντα και μπορούν έτσι να παράγουν νέο πλαστικό βλέπετε ένα κομματάκι πλαστικό το οποίο προέρχεται ακριβώς από τα πολυμερισμένα πλαστικά που επεξεργάζεται η μονάδα καθαρισμού υδάτων των Βρυξελών. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στα πλαίσια της λεγόμενης κυκλικής οικονομικής αντίληψης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε την σωστή τεχνολογία έτσι ώστε αυτά τα βιοδιασπόμενα υλικά, οι σακούλες οι βιοδιασπόμενες να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου στην παραγωγή και σκληρού πλαστικού, έπιπλα, καλάθια, χρήστων κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι στο κείμενό μας μπορούμε εμείς να κινητοποιήσουμε προς την καλύτερη έρευνα και την καινοτομία. Θα πρέπει επίσης να στείλουμε και ένα ισχυρό μήνυμα στις γειτονικές μας χώρες. Πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει το σύνολο της διεθνούς κοινότητας να ευαισθητοποιηθεί. Ξέρετε ότι σήμερα 800.000 ε, τόνους ε, πλαστικές σακούλες μαζεύουμε από ε, τους ωκεανούς και ξέρετε ότι στον Ειρηνικό ωκεανό τεράστιες εκτάσεις με πλαστικές σακούλες απαγορεύουν στα πλοία να τις διαπεράσουν. Είναι σημαντικό λοιπόν να τις διαπλέψουν, να ζητήσουμε από τη διεθνή κοινότητα να ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση και συγχαίρω την εισηγήτρια για μιας πρώτης ποιότητας προσπάθεια. Θα και εγώ να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια δεν νομίζω ότι... και, να... στηρίζω τις εισηγήσεις της. <clears throat> δεν νομίζω ότι στο θέμα της πλαστικής σακούλας μπορεί να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι μετά από όλη τη ζημιά που έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μέτρο που μπορεί να είναι ε, εκτός ε, των ε, σωστών διαστάσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του τρομερού φαινομένου της μόλυνσης από πλαστική σακούλα. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω βέβαια και με αυτά που είπε ο Κάρλος Λούτερ για το θέμα των βιοδιασπαζόμενων και κλείνω με ένα σχόλιο. Αναφέρθηκε και ο Κάρλ Χάνις Φλόρενς για, την, για το θέμα της, της καύσης των σκουπιδιών και αν και το EPP είναι σύμφωνο, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να δούμε το θέμα μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον έλεγχο της διαδικασίας καύση σκουπιδιών, που απειλεί να κλειδώσει, να υποχρεώσει τα πολλά κράτη-μέλη που το εφαρμόζουν να μείνουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα ε, ανακύκλωσης. Ε, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που αυτή η Επιτροπή πρέπει να το κοιτάξει με πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα κλείνοντας να δώσω το λόγο άλλη μια φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θα θέλατε σύντομα, ή θα έχουμε πρόβλημα και με το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα. Uh, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω κάποιες από τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Πρώτα απ' όλα, ο απότερος στόχος της πρότασης, ο βασικός της στόχος είναι η πρόληψη των αποβλήτων, είπαμε την ε, αρχή της ιεραρχίας. Προτού περάσουμε ε, στο θέμα της μεταχείρισης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης, της καύσης, αποτέφρωσης και κουλπού, θα πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή, τη χρήση των, της σακούλας, ώστε να μην δημιουργούνται τόσο πολλά απόβλητα. Αυτός είναι ο αρχικός στόχος της πρότασης, πρόληψη. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το άρθρο 4 της Οδηγίας για τις Συσκευασίε. Εκεί μιλάμε για πρόληψη. Ε, φυσικά, ε, στο πεδίο καλύπτεται και το θέμα της ανακύκλωσης ε, των υπολείπων των αποβλήτων και προσπάθειες που έχουν γίνει σε κάποια κράτη-μέλη δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Για το πεδίο εφαρμογής και πάλι μιλάμε για όλες ε, τις ε, ε, ελαφριές σακούλες κάτω από τα 50 microns, δηλαδή καλύπτουμε τις πολύ λεπτές. Η συγγήτρια θεωρεί ότι αποκλείονται αυτές και υιοθετεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, διότι προτείνει, αντιπροτείνει μάλλον, ευρωπαϊκό στόχο. Εμείς πάλι όχι. Γι' αυτό και στη δική μας προσέγγιση καλύπτουμε ολόκληρο το φάσμα των ελαφ... από τα 50 μάικρον και κάτω για όλες αυτές τις πλαστικές σακούλες θα πρέπει να τεθούν εθνικοί στόχοι μείωσης της χρήσης. Όταν μιλάμε για λεπτές, ε, λιγότερο λεπτές βιοδιασπόμενες, ε, μη βιοδιασπόμενες, πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο να μειωθεί η χρήση όλου του φάσματος. Υπάρχουν και κάποια πιο οριζόντια ζητήματα, πλαστικά απόβλητα ή και πέραν αυτού το θέμα των αποβλήτων ε, Οριστή συλλογή βιοδιασπόμενων είναι ζητήματα που πρέπει να πραγματευτούμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και όχι ε, σε αυτό της συγκεκριμένη πρότασης. Ε, ελπίζουμε ε, του χρόνου όταν θα προτείνουμε αναθεώρηση της οδηγίας για τη συσκευασία και για την ανακύκλωση θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα ανταποκρινόμενοι ε, και ε, στο feedback στις ε, πληροφορίες που ζητήσαμε για το θέμα των πλαστικών αποβλήτων. Σίγουρα δεν είναι το θέμα μας σήμερα. Για το συγκεκριμένο εργαλείο δεν λέει η πρότασή μας ότι πρέπει να προτείνουμε απαγόρευση. Το, τα κράτη-μέλη θα πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το προσφορότερο μέσο χρησιμοποιώντας οικονομικά εργαλεία περιορισμούς στην αγορά ε, κατά το δοκούν θα προτείνει κάθε κράτος μέλος μέτρα για τη μείωση. Φυσικά υπάρχει το θέμα της ε, παιδείας, ε, της ευαισθητοποίησης. Υπάρχουν και τέτοια στοιχεία στην πρότασή μας. υπάρχουν και δεδομένα για την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς του καταναλωτή. Ε, χίλιες πλαστικές ε, σακούλες αν αποσυρθούν από την αγορά τότε αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν άλλου είδους σακούλες, ε, πλαστικές, ε, χάρτινες και άλλων ειδών. Δηλαδή για κάθε χίλιες τέτοιες ε, σακούλες ε, ε, αν αποσυρθούν από την αγορά αντικαθίστανται από 400 σακούλες άλλου είδους κερδίζουμε περίπου 600 σακούλες βάσει των εκτιμήσεών μας. Η αξιολόγησή μας επίσης εξετάζει τον αντίκτυπο στην βιομηχανία για να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Και πάλι βασιστήκαμε στα δεδομένα που έχουμε. Πρέπει να βασιστούμε ε, στη βιομηχανία για τα στοιχεία των αριθμών των θέσεων απασχόλησης, των αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο και εν γέννη κρίνουμε ότι ω προ ε, τα περιβαλλοντικά ωφέλη είναι σχετικά περιορισμένο ο αντίκτυπος ε, της εφαρμογής της πρότασή μα. Για την νομική βάση βασιζόμαστε στο άρθρο 114 ε, επειδή και η αρχική μας πρόταση ε, δραζόταν στην διανομική βάση, το άρθρο 18 της ε, τρέχουσας οδηγίας για την συσκευασία που ουσιαστικά ασχολείται με τα ζητήματα εσωτερικής αγοράς, Ε, και πιστεύουμε ότι η τροποποίηση αυτού του άρθρου πρέπει να βασίζεται επίση στο άρθρο 114. Θέλουμε να υπάρχει συνοχή σε σχέση με τη νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική οδηγία. Και να χρησιμοποιηθεί η ίδια και για την αναθεώρηση. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτήν την νομική βάση. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα σχόλια. Αν τυχόν παρέλειψα κάτι, με τα χαρά να επανέλθω. Να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα... Ναι, ναι, ναι, ήσυχα, ήσυχα. Η συγγετρία έχει το λόγο για να κάνει τα καταληκτικά της σχόλια και να απαντήσει στις ερωτήσεις και να κάνει διάφορες παρατηρήσεις. Η κυρία Όκεν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια και ακούσαμε τόσες πολλές γλώσσες, να μην χρησιμοποιήσω και εγώ τα αγγλικά. Απαντώντας, καταρχάς να απαντήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιστικό όταν μας λέτε ότι εμείς καλύπτουμε όλες τις ε, σακούλες και καλούμε για μείωση όλων των ειδών σακούλα. Χαίρομαι, αλλά δεν έχετε ούτε κάποιο μέσο να προτείνετε, ούτε κάποιο στόχο, μόνο καλέ συστάσεις κάνετε. Άρα, ανυπομονώ να λάβω καλά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Μέρκη, νομίζω, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική ε, λύση για τη συσκευασία του ψαριού. Και ανυπομονώ, γιατί όλα αυτά θα ήθελα να τα συμπεριλάβω να συμπεριλάβω, θα ήθελα μάλλον και τι πολύ ελαφριές σακούλες. Ε, ναι, κύριε Γερμπράντη, εξαιρούνται μεν, αλλά δεν είναι για το κρέα. Εκεί λέμε και περιλαμβάνονται στην πρότασή μου, η πρόταση για τη μείωση. Αλλά δεν τύφεται ειδικό στόχο. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν έχω πρόβλημα για να βρούμε έναν τρόπο μόνο και μόνο να επιλύσουμε αυτό το πολύ βασικό, πρακτικό ζήτημα, το οποίο, για να είμαστε ειλικρινεί, αν ω Επιτροπή λέμε ότι «Α, ναι, θέλουμε καλύτερο κόσμο, θέλουμε να τα μειώσουμε όλα αυτά», το μόνο που έχουμε να σας προτείνουμε όμως είναι «Α, ας τα βελτιώσουμε όλα, χωρίς συγκεκριμένου στόχου. μία ε, απάντηση στην κρίστα. Δεν προτείνουμε απαγόρευση. Προτείνουμε 80% μείωση της μέσης κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός όταν πολλοί λένε ότι άμα τιμωρούμε την τάδε και την συμπεριφορά. Ε, όχι, δεν είναι τιμωρία όταν ε, καλούμε να πατάξουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα και στη Δανία νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα προέρχονται και από τη Δανία. Παρά το γεγονός ότι είμαστε ενδεχομένω οι πιο καλοί μεταξύ των υπόλοιπων ομοτήμων και είμαστε βέβαιοι, είμαι βέβαιη ότι η έκθεση θα είναι καλή. Αν σημειωθούν συγκεκριμένα βήματα. Τώρα, η αναφορά στη συγκεκριμένη μελέτη αντικτύπου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου προκαλεί έκπληξη. Άμα έχετε μια τόσο καλή μελέτη. Μα γιατί με τη χρησιμοποιείτε. Δεν είναι ωραίο. Και νομίζω ότι πάει χαμένη καλή δουλειά αφού δεν τη χρησιμοποιείτε. Να προσπαθήσουμε να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Όταν την είχατε πετάξει λοιπόν στα σκουπίδια, εμείς την ε, βγάλαμε και την επαναχρησιμοποιήσαμε. Θα κάνουμε εμείς ε, λοιπόν αυτή την παρακολούθηση της καλής αυτής της δουλειάς, μιας και με την κάνετε εσείς. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω γιατί νομίζω πολλά καλύψαμε στη σημερινή συζήτηση. Αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια για την βιοδιάσπαση και για την απαγόρευση. Αυτό αναφέρθηκε στην έκθεση της Επιτροπής. Δεν το αναφέρουμε εμείς εδώ. Αν δουλεύουμε με βιοδιασπόμενες σακούλες, θα πρέπει να έχουμε πολύ σαφείς όρους το θέμα δεν είναι μόνο η συλλογή των βιοδιασπόμενων ε, τέτοιων ε, σακούλων, αλλά και διάφορα είδη άλλα βιοδιασπόμενου, βιοδιασπόμενων απορριμμάτων, αποβλήτων. Μόνο όμως αφού είναι βιοδιασπόμενες. Μίλησα για τις ε, πολύ ελαφριές αυτές σακούλες. Τι άλλο ήθελα να τονίσω, κλείνοντας. Χαίρομαι τόσο πολύ, χαίρομαι ιδιαίτερος που από τον Καρλ Χάινς ε, Φλόρενς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σαφές το μήνυμα ότι το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι η πρόληψη. Η πρόληψη όχι με φανταστικούς τρόπους ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση της πλαστικής σακούλας είναι σχεδόν αδύνατη από όσο γνωρίζω. Ακόμα και αν υπάρχει ε, πολύ καλό σύστημα συλλογής, δεν υπάρχει ουσία τόσο πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να ανακυκλωθούν οι πλαστικές σακούλες. Είναι πολύ πενιχρό το αποτέλεσμα τελικά. Αλλά μία σακούλα που περιφέρεται στο περιβάλλον έτσι και είναι πολύ επιβλαβής για το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν η πρόληψη είναι η λέξη κλειδί και πραγματικά είναι φρικτό να βλέπουμε τέτοια μόλυνση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό λοιπόν το σκέλος της πρόληψης θα ήθελα να σας διαβάσω αυτό που αναφέρεται στην τροπολογία 3 Και δική μου. Αναφέρεται ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι πολύ χαμηλά παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολη η ανακύκλωση των, της σακούλας, της πλαστικής σακούλας. Επίσης, η ανακύκλωση της πλαστικής σακούλας δεν αναμένεται να φτάσει σε σημαντικά επίπεδα γιατί είναι πολύ λεπτή και ελαφριά και δεν έχει λοιπόν υψηλή αξία ως προς την ανακύκλωση. Είναι επίσης δαπανηρή η μεταφορά τους και η ανακύκλωση της πλαστικής σακούλας λοιπόν δεν επιλύει το πρόβλημα το οποίο προκαλούν και γι' αυτό λοιπόν πρώτος στόχος προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η πρόληψη. Εκ νέου χρήση, ναι. Ανακύκλωση όμως, όχι. Αυτό δεν έχει νόημα να τεθεί επιτάπητος. Νομίζω όμως ότι έτσι έθιξα και απάντησα στις ερωτήσεις που ετέθησαν και προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία για να ολοκληρώσουμε το στομότερο δυνατόν την επεξεργασία της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άουκεν, λέει ο Πρόεδρος. Στις 27 Ιανουαρίου έχουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 12. Όπως είπα σήμερα το πρωί ήδη, μέχρι την Παρασκευή διατίθεται, θα διατίθεται ένα εργαλείο στο διαδίκτυο όπου οι βοηθοί και οι βουλευτές θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό υποδοκιμή. Στις 6 Μαρτίου θα ψηφίσουμε και επιλέξαμε τη δεύτερη ολομέλεια του Απριλίου για να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και έτσι μπορούμε να περάσουμε στην έκθεση του συναδέλφου Σκυλακάκη. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Η έκθεση για τις uh, εκπομπές θαλασσίων μέσων, σκαφών Ελπίζω να προχωρήσει σε μια, με θετική έκβαση, να ολοκληρωθεί η διαδικασία θετικά. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι όπως είπα να καταλήξουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της ε, παρούσης κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε μετά από την ψηφοφορία μας στις 30 του μηνός να έρθουμε σε επαφή με την Ελληνική Προεδρία και να μπορέσουμε να κλείσουμε κατά τη διάρκεια της περίοδου τη διαδικασία. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό, δεν έχουμε δηλαδή πάρα πολύ χρόνο. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια κάποια συμφωνία μετά την Ολομέλεια. Πριν γίνει αυτό βέβαια θα πρέπει να ψηφίσουμε και στη δική μας Επιτροπή. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες συμβιβαστικές προτάσεις και στο εσωτερικό ε, ε, του Κοινοβουλίου μας. Υπάρχουν ορισμένα θέματα κρίσιμα θα έλεγα. Πρώτον, η εμβέλεια. Εμείς εγώ θα ήθελα να διευρύνουμε την εμβέλεια και να συμπεριλάβουμε και τα νοξ, Όπως ξέρετε είναι και τα νοξ ε, ε, αέριο του, του θερμοκηπίου. Δεν ξέρω αν ε, η προσπάθεια που θα γίνει θα είναι θετική ή αρνητική σε σχέση με την προστασία του κλίματος, αλλά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα νοξ. Αυτή είναι η πρόταση την οποία έχω και στις συμβιβαστικές τροπολογίες και σε ό,τι άλλο. Ελπίζω ότι θα διευρύνουμε την εμβέλεια και για το τι σκάφη θα καλύψουμε, να καλύψουμε και τα μικρά σκάφη, μικρού μεγέθους. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει εμείς να ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό άχθος θα έλεγα και να μην συμπεριλάβουμε μέτρα επιβαρυντικά στην προσπάθεια καταμέτρησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα, αλλά δίδοντας αρκετά δημόσια δεδομένα ανακοινώσιμα σε όλους την αγορά έτσι ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Γενικότερα λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε το τι θέλουμε πράγματι να κάνουμε με την ομοθετική αυτή ρύθμιση. Προσπαθούμε να πιέσουμε τον Διεθνή ε, Θαλάσσιο Οργανισμό, το IMO, να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των σκαφών του και να προετοιμαστεί για την εφαρμογή της αρχής ε, αυτός που μολύνει πληρώνει σε όλους τους τόλους ε, στον κόσμο. Υπάρχουν δύο τρόποι να το πετύχει αυτός μακροπρόθεσμα είτε με ένα σφαιρικό τέλος, ένα συνολικό σφαιρικό τέλος και αυτό θα πρέπει να στοχεύσουμε νομίζω. Ένα τέτοιο τέλος νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να εφαρμοστεί, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε στο μέλλον. Πάντως πρέπει να εφαρμόσουμε την βασική αυτή αρχή και για τις θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο εμπόριο. Και το θέμα δεν είναι μόνο να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, που είναι ένας γενικότερος και παράλληλος στόχος. Θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και είναι ένα αρκετά καλό κίνητρο αλλά νομίζω ότι βασικός στόχος είναι η εφαρμογή της αρχής όποιος μολύνει πληρώνει. Και για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορικές θα πρέπει να πληρώνουν αυτό το οποίο οφείλουν για τις εκπομπές ε, καυσαερίων στην ατμόσφαιρα. Ελπίζω λοιπόν επί τη βάση αυτών των στοιχείων να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη και κατά τη διάρκεια της ψήφου. Πολλές από τις συμβιβαστικές α, τις έχουμε πετύχει, σε κάποιους άλλους τομείς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα πρέπει να το λύσουμε αυτό μέσω της ψηφοφορίας. Μετά την ψηφοφορία πάντως ελπίζω να προχωρήσουμε στους τριμερείς διαλόγους και να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα μέσω μιας συμφωνίας κατά τη διάρκεια της παρούσης κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτή είναι η ελπίδα μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης και όλους όσους εργάστηκαν σκληρά για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε κάποιο δρόμο να διανύσουμε ακόμα μέχρι την ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα. Christopher Fjellner hat Sorry, zu Sozial I'm kind of zu den Sozialdemokraten. Yeah, I slid to the wrong part. Ε, ο Christopher Fjellner, ναι, ζητώ συγγνώμη και πήγα από τη λάθος πλευρά. Και δεν νιώθω και άνετα σε αυτή τη θέση, οφείλω να ομολογήσω, όμως νιώθω άνετα με αυτό το ζήτημα. Anyhow, let's get to business. Uh, for... Τέλος πάντων, δεν μπορώ, λέω εξ αρχής, ε, να μείνω μέχρι το τέλο της συζήτηση, γιατί πρέπει να πάρω νωρί την πτήση μου αλλά ε, ήθελα να πω ότι στο πλαίσιο της συζήτησης είναι σημαντικό να πούμε ότι ε, για τις οι θαλάσσιες μεταφορές ε, είναι και αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον σε σχέση με τα, τους άλλους τρόπους μεταφοράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα διότι οι άλλοι τρόποι μεταφοράς είναι πολύ χακοί. Οπότε δεν θα έπρεπε να κάνουμε οτιδήποτε είναι αντιπαραγωγικό. Ό,τι και αν αποφασίσουμε ο στόχος μας θα πρέπει να είναι με αυτόν τον κανονισμό να βρούμε μια ε, λύση ικανοποιητική ε, παγκόσμιας κλίμακας. Εγώ θεωρώ ότι είναι, ε, καλά, είναι ισορροπημένη και ικανοποιητική η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συμβαστικές που επεξεργάζεται ο κύριος Κυλακάκης και τα αποτελέσματα της δουλειάς των σκιωδών επίσης με ικανοποιούν. Δύο ζητήματα ήθελα μόνο να θέσω υπόψη σας ε, για την ολική ε, χωρητικότητα και το όριο. 500 ε, GT θέτει ως όριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι πρέπει να εξαιρεθούν τα μικρότερα σκάφη διότι επισύρει αυτό υπερβολικό διοικητικό άχθος. Αυτό είναι το επιχείρημα της Επιτροπής. Πιστεύω ότι δίκιο έχουν σε σχέση με τα ωφέλη προς το περιβάλλον, αν τελικά καλύψουμε και αυτά τα σκάφη, αν καλυφθούν και ε, τα όσα υπερβαίνουν ε, τα 500 GT, τότε αυτό σημαίνει ότι καλύπτουμε 50% του στόλου και ε, το 91% των εκπομπών. Ορισμένοι θεώρησαν ότι έπρεπε να τεθεί το όριο στα 400 GT και ε, καλύπτοντας έτσι 91% του στόλου και 99% των εκπομπών. Όμως ε, για να συμβεί αυτό, για να περάσουμε από το 57% στο 91% ε, είναι ένα ε, τεράστιο βήμα για να κερδίσουμε ε, μόνο κάποιες ποσοστιαίες μονάδες ε, για τις εκπομπές. Αξίζουν οι επενδύσεις, είναι λογικό να κάνουμε τέτοια επένδυση. Και πάλι Ξαναλέω, σε σχέση με τον αρχικό μας στόχο και τις αρχικές μας επιδιώξεις, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ήδη συλλεχθέντα δεδομένα και να ασχοληθούμε συγκεκριμένα με τις εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα, διότι ξέρουμε δύο μεγάλοι ρηπαίνοντες ε, είναι το θείο και το διοξίδιο του άνθρακα. Με την κυρία Χάση ε, ε, ασχολούμαστε με το θείο στα πλαίσια της αντίστοιχης οδηγίας και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το διοξίδιο του άνθρακα. Γίνονται διάφορες απόπειρες διεύρυνσης του πεδίου και ο κύριος Χιλακάκης μας μίλησε για τα διοξίδια του αζότου και ε, τα, τα και πιστεύω ότι ε, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα συμφωνίας με το Συμβούλιο, γιατί αυτό είναι βασικός μας στόχος. Και δεύτερον, θα έπρεπε να ε, διευκολύνουμε την επίτευξη ε, του συνολικού μας στόχου, δηλαδή να έχουμε συμφωνία σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, IMO. Αυτά είναι τα δύο σημεία που θα έπρεπε να ε, ε, ξανασκεφτούν οι συνάδελφοι. Να περάσουμε δηλαδή στα 400 ε, GT. Έκανε λάθος ο μιλητής και μίλησε για gigatons που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό ε, και να ε, μην ασχοληθούμε με τις, ε, δι, με, με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν, είναι, δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε όλα με μία πρόταση. Ευχαριστώ και πάλι ο Κρήτον Σένης από αριστερά. Ε, I would like Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τις προσπάθειες που έκανε για συμβιβασμό και για την προσπάθεια να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα για τη συμφωνία αυτή στα πλαίσια της θητείας αυτής. Συζητήσαμε στην ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, την διαδικασία για εξέβρεση συμβιβασμού. Να κοιτάξουμε όμω τι τροπολογίε τις συγκεκριμένε τι οποίε θα υποστηρίξουμε και στον κατάλογο ψηφοφορία πέρα από το συμβιβασμό. Για μα. υποστηρίζουμε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ε, και συμπεριλαμβανομένων των των οξυδίων του αζότου, για να χαμηλώσουμε τώρα το όριο για τα σκάφη από τα 500 από 5.400 από 500 σε 400, ε, αυτό είναι θέμα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογή, αλλά μπορεί να είναι και θέμα όπου το ΕΛΚ συχνά στην ομοθεσία έχει αυξήσει τη διαρροή άνθρακα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης υποβάλαμε τροπολογίες και ζητήσαμε να καταργηθεί σταδιακά σε πέντε έτη η μέθοδο που είναι λιγότερο εξελιγμένη της παρακολούθησης του διοξιδίου του άνθρακα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό προκειμένου σταδιακά να αυξηθεί και η ακρίβεια της παρακολούθησής μας. Κάτι άλλο. Το θέμα των βιοκαυσίμων, πολύ γνωστό εδώ στην αίθουσά μας. Προτείνουμε στο παράδειγμα 1α τα βιοκαύσιμα να εξισωθούν με τα συμβατικά καύσιμα όσο δεν υπάρχει μια αξία προορισμένη, γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με το σύστημα αυτοεξοικονόμησης. Ή θα είμαστε ακριβείς ή αλλιώς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν τα βιοκαύσιμα. Όπως έχει διακαυθεί η συζήτηση στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, ένα βασικό ζήτημα είναι η αλλιως δεν μπορουν να συμπεριληφθουν τα βιοκαυσιμα οπως εχει διεκαθει η αποδοτικότητα και τα στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να προσμετρήσουμε με ακριβή τρόπο την αποτελεσματικότητα των σκαφών αυτών, την αποδοτικότητα των σκαφών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και για μας και γενικότερα. Και γιατί? Γιατί η καταμέτρηση, η προσμέτρηση της αποδοτικότητας δημιουργεί ένα σαφές πρότυπο για την δευτερογενή αγορά. Όταν ο κόσμος πουλάει για παράδειγμα τα σκάφη αυτά εφόσον γνωρίζει ο κόσμος τι αγοράζει, θα θέσει προτεραιότητες και θα προτιμήσει ασφαλώς τα πλέον αποτελεσματικά, τα πλέον αποδοτικά. Αυτό λοιπόν ε, ε, ευνοεί την επένδυση σε αποδοτικά σκάφη. Αυτό το θέλουμε σε όλη τη νομοθεσία, το θέλουμε και εδώ. Και αυτό λοιπόν συζητιέται στα πλαίσια του IMO. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλωσορίσω μία πρώην συνάδελφο, την Ντόρετ Κόρμπεϊ. Ντόρετ, hartelijk welcome. Καλώ ήρθε, Ντορέτ, στην Επιτροπή μα. Επόμενο ομιλητής, η κυρία Σατουχάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για τις προσπάθειες που έκανε ε, για να καταλήξει ε, σε συνεργασία με άλλες πολιτικές ομάδες σε μια συμβαστική λύση. Υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία ε, που μπορούμε να υποστηρίξουμε στην πρόταση του εισηγητή και η πράσινη το ίδιο. Τα προς τα νόξ, ας πούμε, τα οξύδια του αζότου μας βρίσκουν σύμφωνος. Κάλυψη των αερίων του θερμοκηπίου γενικότερα και όχι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Μείωση του ορίου στα 400 GT αλλά δεν μπορώ να ε, υποστηρίξω τα πάντα. Ε, Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιδιώξουμε την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των θαλασσίων μεταφορών και να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των πελατών της ναυτιλίας, ώστε να έχουν στοιχεία στη διάθεσή τους και να επιλέγουν ε, φορείς εκμετάλλευσης που ενεργειακά είναι πιο αποτελεσματικοί. Ε, από πού απορρέει αυτή η πρόταση, το ε, θυμηθούμε διότι έχουμε απομακρυνθεί ε, αργά αλλά σταθερά από την αρχική πρόθεση του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο κίνησε τη διαδικασία το 2008 στα πλαίσια του πακέτου για την κλιματική αλλαγή και αυτό εξετάζαμε τότε και ζητήσαμε ε, ότι όλη η διεθνής ναυτιλία θα πρέπει να εφαρμόζει μέτρα για τις κλιματικές αλλαγές ε, και ζητήσαμε για την οδηγία ETS ε, και για την ε, απόφαση για τον επιμερισμό των προσπαθειών να αναφέρουν ότι για το 2011 δεν υπάρχει κανένα μέτρο, κανόνας του IMO, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμού και ως εκ τούτου θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τα δικά της μέτρα, είτε ε, ε, καλύπτοντας τη διεθνή ναυτιλία μέσα στο σύστημα δικαιωμάτων εκπομπής είτε καλύπτοντας τα καυσαέρια ε, που, των πλοίων απλώς. Λοιπόν, αυτή η πρόταση ε, υπολείπεται του αρχικού μας ε, στόχου που θέσαμε, ξαναλέω, προπενταετίας απογοητεύτηκα που υπάρχουν τόσοι πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο που θέλουν να αποδυναμώσουν έτσι περαιτέρω αυτή την ήδη αδύναμη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά, να μην ξεχνούμε ότι ε, στην παγκόσμια αγορά ε, το κομμάτι των ε, αερίων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη διεθνή ναυτιλία βρίσκεται στα ίδια επίπεδα όπως ε, και στην αεροπορία ε, περίπου ε, και έχουν τον ίδιο ρυθμό αύξησης. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε προσπάθειες για να μειώσουμε τις εκπομπές και στους δύο αυτούς τομείς, την ναυτιλία και την αεροπορία, αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι δύο τομείς μας τρώνε και καταλαμβάνουν το περιθώριο ελιγμών που έχουμε ε, για άλλους τομείς. Ε, το lobbying ε, που γίνεται δείχνει ιδιαίτερη συνέπεια. Δηλαδή, στις, στους τομείς βιομηχανίας με μεγάλη ένταση ενέργειας γίνεται εντατικό lobbying υπέρ των θαλασσίων μεταφορών για την αστυλία παραδείγματος χάρη για να συμπεριληφθούν μόνο οι εκπομπές ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα. Ξαναλέω, ε, απευθύνω έκκληση μάλλον, να μην αποδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός από την δεξιά πτέρυγα, ο δεξιός Μάρτιν. Παρακαλώ Μάρτιν from your new birth alongside the forces of darkness over there. It's good to see you back on the right side. Χαίρομαι που σας βλέπω από τη σωστή πλευρά μετά από την πλευρά του σκότους. Λοιπόν, εγώ αντίθετα ε, από τους πρασίνους θεωρώ ότι είναι θετικά τα στοιχεία που περιλαμβάνει η πρόταση αυτή. Είναι μια πραγματιστική πρόταση, μια έλογη πρόταση, μια δίκαιη πρόταση που αφορά επίσης και ε, ε, τα επιβατικά πλοία τα οποία κανονικά υπό τις προηγούμενες προτάσεις θα είχαν φυγεί ιδιαίτερα. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι σε σχέση με τον κανονισμό αυτό. Είναι το πρώτο βήμα αυτό τον οποίο κάνουμε και όπως λέγει και το όνομα θα πρέπει να παραμείνουμε στο θέμα της, του υπολογισμού αξιολόγησης και αναφοράς θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θα πρέπει ίσως να συμπεριλάβουμε και άλλα αέρια του θερμοκηπίου, αφού όμως αναλύσουμε το κόστος και τα ωφέλη μιας τέτοιας μεθόδου και τεκμηριώσουμε την επιλογή αυτή. Και γι' αυτό δεν εγώ εγκρίνω τη συμπερίληψη των αερίων NOx. Ε, υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι για τον υπολογισμό των εκπομπών. Θα πρέπει φυσικά και προς όφελος της βιομηχανίας αυτής να χρησιμοποιεί το λιγότερο δυνατό καύσιμο και δεν θα πρέπει να επιλέξουμε μόνο τις δύο πιο ακριβές. χωρίς να επιβαρύνουμε φυσικά ιδιαίτερα τους πλειοκτήτες και ταυτόχρονα να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Άνω των 5.000 τόνων μικτού βάρους, όπως ακριβώς ε, είπατε, αυτά τα μεγάλα σκάφη αποτελούν το 90% της συνολικής μόλυνσης. Νομίζω το να πάμε από τους 5.000 στα 400, στους 400 τόνους, αυτό σημαίνει υπερβολική γραφειοκρατία για τους ε, πλειοκτήτες αυτών των μικρών σκαφών με ελάχιστες ε, ε, εκπομπές να καλύπτονται επιπλέον μόνο 10%. και ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιηθούν οι δύο πιο ακριβές μέθοδοι για τον υπολογισμό των εκπομπών. Ευχαριστώ Μάρτιν. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ ή εκπρόσωπος. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους κοιόδης για τις πολύ καλές τους προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρξει μια ικανοποιητική συμβιβαστική λύση με επικοδομητικά αποτελέσματα σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε με τις εκκρεμότητες αλλά να προσπαθήσουμε να τις ιεραρχήσουμε εμείς τουλάχιστον στην Επιτροπή με διαφορετικό τρόπο και σε σχέση με την εμβέλεια και σε σχέση με τη διαφάνεια βασικοί στόχοι of της πρότασης MRV είναι μεγαλύτερη διαφάνεια και αλλαγή των ε, συμπεριφορών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα έχει πάντα σαν στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εάν δεν συμπεριλάβουμε ορισμένες πληροφορίες όπως τα εμπορεύματα, τα μεταφερόμενα στα πλαίσια του MRV, και αν δεν καταστήσουμε τις πληροφορίες αυτές ευρύτερα γνωστές, τότε δεν θα προκαλέσουμε τις αλλαγές αυτές τις οποίες επιθυμούμε και φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε. Σίγουρα λοιπόν ένα ισχυρό MRV είναι το θεμέλιο για η αδίποτε περαιτέρω δράση έτσι ώστε να προκαλέσουμε τα αποτελέσματα τα οποία εμείς θεωρούμε σωστά ε, στην αξιολογήσή μας. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι πάρα πολύ εύκολα να διασφαλίσουμε απλά τη διαφάνεια της ενημέρωσης, ε, κάτι το οποίο είναι όχι δευτερεύον αλλά είναι ένα μεθοδολογικό τμήμα της βασικής διαδικασίας. Έχουν γίνει αρκετές εξηγήσει από πλευράς μας γιατί δεν είχαμε συμπεριλάβει τα νόξο στην πρότασή μας. Οι τεχνολογίες για την καταμέτρηση των νόξο τεχνικά δεν είναι απόλυτα διαθέσιμες. Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι με κάποια θετικά αποτελέσματα. αλλά οι εκτιμήσεις για το κόστος των επενδύσεων για την προσμέτρηση είναι σχεδόν 100.000 ευρώ ανά σκάφος και όταν μιλάμε για δεκάδες, ε, εκατοντάδες και χιλιάδες ε, σκάφη τότε καταλαβαίνετε ότι ε, αυτό δεν είναι εφικτό και σε της άλλης δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε και τη διαδικασία. Σχετικά με το κατώτατο όριο αναφερθήκατε στο θέμα του τονάζ Από τη μία έχουμε την αύξηση του ποσοστού των εκπομπών και από την άλλη την αύξηση του αριθμού των πλοίων. Δεν θα σταθώ σε αυτά. Αν μειώσουμε το κατώτατο όριο, σε αυτή την περίπτωση θα συμπεριλάβουμε φυσικά και πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ περισσότερο διοικητικό βάρος να αντιμετωπίσουν γραφειοκρατικό κτλ. Ε, βασικός μας στόχος θα πρέπει να συνοδεύεται με πραγματισμό. Κάποια μικρά σχόλια για αυτά τα οποία ακούστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής και τους κοιόδης εισηγητές. Οι μέθοδοι καταμέτρησης, εμείς προτείναμε τέσσερις μεθόδους, θεωρούμε ότι αυτό είναι αναλογικά σωστό και διοικητικά απλό οι μεθοδολογίες υπάρχουν ήδη εν πολλής και θέλουμε εμείς να διασφαλίσουμε την ευκολία εφαρμογής τους από πλευράς των χρηστών. Έχουν γίνει και ορισμένες προτάσεις για το χρονοδιάγραμμα και εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι αν και το 2018 φαίνεται ότι είναι μακριά, Υπάρχουν ε, και διάφορα νομικά μέτρα, εφαρμοστικές πράξεις και τεχνικές ε, προπαρασκευές που είναι απαραίτητες και για τα κράτη-μέλη και για την συγκεκριμένη ε, επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτά. Πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ο εισηγητής έχει το λόγο πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις για τον συγκεκριμένο κανονισμό. Ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποιες καλές συμβιβαστικές λύσεις στο τέλος. Για την ενεργειακή αποδοτικότητα θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν τεράστια κίνητρα για την ναυτιλιακή βιομηχανία. Ξοδεύουν το 2 τρίτα του κόστους της λειτουργίας τους είναι τα καύσιμα μπορούν φυσικά να εκμεταλλευτούν την νέα κατάσταση εφόσον υπάρχουν περισσότερα δεδομένα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τα δεδομένα τα οποία ελείπουν σήμερα για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα ενεργειακά. Το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας στην αυτιλιακή δραστηριότητα είναι περίπλοκο πράγμα, εμπλέκει πάρα πολλά πράγματα, όπως τα ρεύματα, την καθαριότητα του κήτους του σκάφους, το βήμα των προπελών που κινούν το σκάφος, ε, καιρικές συνθήκες φυσικά, ο άνεμος κτλ. Ε, δεν υπάρχει δηλαδή ένα μαγικό ραβδί δεδομένων τα οποία θα περιμένει ο κόσμος να χρησιμοποιήσει όταν τα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Δεν είναι αυτή η βάση του κανονισμού. Η βάση του κανονισμού είναι κάτι το πάρα πολύ απλό. Τα σκάφη εκπέμπουν. Ε, αυτό είναι αρνητικό για το κλίμα. Στην παρούσα στιγμή δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει εμείς να καταμετρήσουμε τις εκπομπές ανασκάφος έτσι ώστε να εφαρμόσουμε σωστά τις αρχές τις οποίες ανέφερα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι τα μικρά σκάφη γενικότερα δεν θα πρέπει να πληρώσουν για τη μόλυνση, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Όλοι θα πρέπει να πληρώνουν εφόσον μολύνουν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα μικρότερα σκάφη. Γνωρίζουμε ότι τα μεγάλα σκάφη φυσικά μπορούν να είναι πιο αποδοτικά στον τομέα της κατανάλωσης και δεν θέλουμε εμείς να προχωρήσουμε σε αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις και να πιέσουμε ε, τα μικρά σκάφη ε, σε μικρότερη ενεργειακή αποδοτικότητα μέσω της εξαίρεσής τους. Λοιπόν, θα πρέπει εμείς να ε, δώσουμε τη δυνατότητα ενός εύκολου MRV, εφόσον το κάνουμε αυτό τώρα, θα πιέσουμε το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ε, σε ευκολότερες και γρηγορότερες λύσεις. Πρέπει να γίνει σε αυτό το κοινοβούλιο να ολοκληρωθεί η προσπάθεια γιατί αυτό σημαίνει τουλάχιστον μια διαφορά χρονική ενός έτους. Λοιπόν, ελπίζω να τα καταφέρουμε στον λίγο χρόνο που έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ κύριε και κύριοι, έτσι ολοκληρώσαμε την, ε, την συζήτηση. Θα ψηφίσουμε στην ε, ε, Επιτροπή μας στις 30 Ιανουαρίου και έχουμε λοιπόν τον την τελευταία ευκαιρία να το ολοκληρώσουμε αυτό και σε πρώτη ανάγνωση. 30 Ιανουαρίου για τις ε, τροπολογίες. Και τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι το σημείο 23. Η κυρία Σάτου Χάση είναι εδώ. Πρόκειται για την εφαρμογή του άρθρου 7α τη Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων. το έχουμε μια προφορική ερώτηση της κυρία Σατουχάση. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Σατουχάση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σήμερα δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της για το πακέτο για την ποιότητα των καυσίμων. Ε, από το πακέτο 2020 μόνο η ποιότητα των καυσίμων ε, δεν έχει εφαρμοστεί παρότι έχει κλείσει πενταετία σχεδόν, ε, μάλλον έχει ήδη κλείσει πενταετία από την θέσπιση της νομοθεσίας. Υπάρχει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, πέρσι έγινε και αξιολόγηση αντικτύπου, όμως δεν έχουν δημοσιευθεί τα συμπεράσματα τα εφαρμοστικά μέτρα έπρεπε να είχαν θεσπιστεί ε, πριν από τρία χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2011. Για το πακέτο 2020 τίθενται δύο ζητήματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης αντικτύπου με αποδέκτες στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως διότι ε, σε σχέση με το εκτιμόμενο κόστος για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι ε, βάσει της μελέτης δεν υπάρχει σημαντικό ε, γραφειοκρατικό άχθος ούτε και σημαντικό κόστος με την εφαρμογή της πρότασης. Δεύτερον, πότε σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει την αναθεωρημένη πρόταση περί εφαρμογής των ε, μέτρων. Τρίτη ερώτηση που σχετίζεται με αυτά που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή είναι η εξής. είπε η Επιτροπή μετά το 2020 δεν θα έχουμε συγκεκριμένους στόχους για την οδηγία ποιότητας των καυσίμων. Αυτό ε, μακροτηριάζει τη, την πρόταση. Αυτό δεν συνδέεται ακριβώς με την αρχική μου ερώτηση, αλλά είναι ε, για να συναφές ζήτημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μόνο εγώ ενδιαφέρομαι για το λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κρίνει σκόπιμο να θέσει νέους στόχους μετά το 2020 για την οδηγία ποιότητας των καυσίμων. Αυξάνονται οι εκπομπές ε, στις μεταφορές, ενώ οι εκπομπές σε άλλους τομείς μειώνονται. Ε, και ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να οι μεταφορές να γίνουν πρωταθλητές ε, ως προς το σύνολο των εκπομπών τους μετά το 2020. Όλοι ξέρουμε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην καναδική πίεση και τις ε, ε, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ένωση και τον Καναδά για τις εμπορικές συναλλαγές. Όμως ε, δεν πρόκειται μόνο για την ε, ε, ασφαλτούχο ε, άμμο και το ασφαλτούχο ε, σχιστολιθικό πετρέλαιο που παράγεται εκεί πρόκειται και για δίζελ σχιστολιστικό αμερικανικό πετρέλαιο που βάσει πληροφοριών που έχω εγώ έχει ακόμη χειρότερο αποτύπωμα οικολογικό από το ασφαλτούχο σχιστολιθικό. Η, Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μη παραδοσιακές, αν θέλετε, ε, πηγές ε, αναδεικνύονται σε προτεραιότητα σήμερα και ε, έχουν αυξανόμενη σημασία. Οπότε για το μέλλον είναι πιο σημαντικό να έχουμε κριτήρια ως προς το οικολογικό αποτύπωμα για τις μεταφορές μας. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε κυρία Μακέβανα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι κατά σύμπτωση που βρίσκομαι εδώ σήμερα, που είναι εδώ από πλευρά της Επιτροπής εκπρόσωπος, γιατί η οδηγία αυτή ε, ενδεχομένως να περάσει στο τελευταίο αυτό κομμάτι. been waiting for donkey's years now. Είναι σύμπτωση που είναι εδώ η μαζί μας σήμερα γιατί που συζητάμε το θέμα αυτό, γιατί σήμερα είναι μια λυπηρή ημέρα για την ευρωπαϊκή πολιτική αλλαγή του κλίματος, γιατί ήταν πολύ αδύναμη και αδιάφορη η δήλωση το 2030 σε ό,τι αφορά τους στόχους. Δεν είναι δεσμευτική η στόχη για τα κράτη-μέλη. Ίσως λοιπόν... Τι θα επινοήσουμε ένα κράτος μέλος για να πούμε ότι κάποιος πέτυχε κάποιους στόχους. Είδαμε τις εκπομπές για την αεροπλοεία και ότι οι στόχοι αποδυναμώθηκαν. Αναρωτιέμαι τελικά όλα αυτά ε, έχουν να κάνουν με την πολιτική για την αλληλεγγύη του κλίματος, ε, με την καναδική πολιτική, με την αμερικανική πολιτική για το θέμα της κλωνοποίησης, το οποίο θα το συζητήσουμε σε άλλη περίσταση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποδυναμώνονται για να ταιριάξουν με τις αμερικάνικες. Για την βιομηχανία αρκτών καυσίμων είναι καλή ημέρα. Έχουν πετύχει πολλοί από τους στόχους τους. Και εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε γνωρίζουν ότι δεν έχει μείνει πολύ καιρό και για το πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν κατηγορώ και την Επίτροπο Έχει πολεμήσει, αγωνιστεί για το θέμα αυτό. Την μπλοκάρουν όμω ε, από πλευρά ε, τη Επιτροπή ή άλλοι Επίτροποι και είναι και πολύ αδύναμη η ηγεσία του Μπαρόσο. Τι θα πούμε λοιπόν από πλευρά τη ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τη σημερινή ημέρα. Πολύ απογοητευτικά τα νέα. Καθίσαμε εδώ, ακούσαμε όλε τι ερωτήσει στην Ολομέλεια και παρόλα αυτά σε κάποια χρόνια θα έχουμε ακόμα α, τέτοια βρώμικα καύσιμα. Γιατί αν όλοι ξέρουν ότι δεν θα επαναληφθούν αυτοί οι στόχοι, ποιος θα τους εφαρμόσει. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε που στον επόμενο κοινοβούλιο. Είναι κρίμα που είναι τόσο λίγοι σήμερα οι συνομιλητές για το θέμα αυτό και είναι λυπηρή αυτή η μέρα. Ντορέτ, πολύ λυπάμαι. Είναι λυπηρή η μέρα σήμερα για την ευρωπαϊκή πολιτική. Χερπερτιάν. Ας ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσω το ερώτημά μου αφού πάρουμε μια κάποια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να ακούσω την απάντησή τους πρώτα. Βεβαίω, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε το κατάλογο των αμελητών Να δώσω το λόγο στον Φιλιππό για να απαντήσει τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Thank you, uh, Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Χάση για τις τρεις ερωτήσεις που θέσατε. Ελπίζω να μπορέσω να μιλήσω λίγο και για την τρίτη ερώτηση, αν και δεν μπορώ να σας δώσω τελική απάντηση. Είναι αλήθεια ότι η διαδικασία είναι μια μακρά διαδικασία, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2009 και όλοι θα είμαστε ιδιαίτερως ευτυχείς να προχωρήσουμε γρήγορα. Είχαμε μία συνάντηση των εμπλεκομένων τον προηγούμενο Απρίλιο, συμμετείχε και το Κοινοβούλιο, μπήκαμε στις λεπτομέρειες του τι θέλουμε να κάνουμε σχετικά με τη μελέτη επιπτώσεων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής συγκεντρώσαμε την προσοχή μας σε κάποια μεθοδολογικά θέματα, μέσα από τα οποία θα προσπαθήσουμε εμείς να καταμετρήσουμε τις προτάσεις και να καταλήξουμε σε έναν μέσο κοινοτικό όρο, έτσι όπως θα ήθελε και η βιομηχανία, Υπάρχουν κάποια επίπεδα τα οποία δίνουν τα κράτη-μέλη. Όλες οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν, είτε οι δυνατότητες από περιοχές όπου υπάρχει παραγωγή από Again, this is technically possible. It's, it's quite difficult, but it's actually possible to, to measure the greenhouse gas emissions from individual oil wells. Σύγκριση, εν πάση περιπτώσει, ε, των διαφόρων ε, ε, τρόπων παραγωγής ενέργειας είτε από σχιστολιθικά πετρώματα είτε από περιοχές με εκτάσεις πίσας κτλ. Το θέμα είναι πόσο θα μπορέσουμε να μειώσουμε το ποσοστό των καυσίμων στο, στις εκπομπές που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Ξέρετε ότι θα υπάρχουν ε, ε, κάποιες παραγωγές ε, και τρόποι παραγωγής οι οποίοι στην Ευρώπη σαν παράδειγμα μπορεί να είναι χαμηλού, χαμηλής περιβαντολογικής επίπλωσης ενώ σε άλλες περιοχές μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη. Βλέπουμε επίσης και τα αέρια τα οποία διαφεύγουν κατά τη διάρκεια της φάσης εξόριξης να μειώνονται τον τελευταίο καιρό και το κόστος αυτό το έχει ήδη αναλάβει η βιομηχανία. Το δεύτερο τμήμα είναι το διοικητικό γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει να ελέγξουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι ε, το διοικητικό κόστος αυτό το έχουμε κρατήσει στο ελάχιστο δυνατόν και αυτό επιβεβαιώνεται και από την έκθεση της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Νομίζω λοιπόν ότι το διοικητικό βάρος δεν είναι όπως είπα πάρα πολύ υψηλό, το παραδέχεται αυτό και η βιομηχανία και το κόστος συμμόρφωσης είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο ε, φοβάται η βιομηχανία ότι θα αναλάβει. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στη μελέτη επιπτώσεων η οποία έχει ολοκληρωθεί εν πολλής και όπως στις περισσότερες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά την έκθεση αυτή διαθέσιμη εφόσον η τελική πρόταση έχει διαμορφωθεί. Δεν έχουμε φτάσει εμείς στην φάση της τελικής πρότασης. Ο Επίτροπος μου, όπως επίσης και πολλοί συνάδελφοι, ασχολούνται με το πακέτο 20-30 τους τελευταίους μήνες. Πολλοί συμφωνούν, πολλοί διαφωνούν με την ανακοίνωση 20-30, αλλά νομίζω ότι μία μείωση 40% ε, είναι, η μείωση των εκπομπών είναι ε, πολύ καλός στόχος. Πολλοί εμπλέκονται λοιπόν στην προσπάθεια αυτή τους τελευταίους μήνες και γι' αυτό ακριβώς ίσως η οδηγία δεν έχει αντιμετωπιστεί με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι θα επιθυμούσαν τον τελευταίο καιρό. Θα επανέλθουμε πάντως στο θέμα στην παρούσα περίοδο δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα στην φάση αυτή σήμερα, αλλά ο Επίτροπός μου θέλει να ολοκληρωθεί η πρόταση αυτή όσο είναι ε, στη, κατά τη διάρκεια της περίοδου ε, ε, που είναι Επίτροπος. Δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν να σας παρουσιάσουμε την πρόταση αυτή κατά τη διάρκεια της δικής σας κοινοβουλευτικής περίοδου. Δυστυχώς Κάνουμε ό,τι μπορούμε, το γρηγορότερο δυνατόν θα γίνει η πρόταση, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σας καταθέσουμε την πρόταση αυτή πριν από την συνεδρίαση του μηνός Απριλίου, την Ολομέλεια την τελευταία. Αυτά και μπράντι. Φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο απογοητευτικά τα πράγματα από ό,τι περίμενα όλα τα επιχειρήματα κατά τις οδηγίες για την ποιότητα των καυσίμων λέτε δεν είναι σημαντικά και σχετικά με το θέμα. Και βάσει την ε, ανάλυση που κάναμε βλέπουμε ε, λέτε, διαψεύδεται διάφορα στοιχεία σε σχέση με το γραφειοκρατικό άχθος, με το κόστος της ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ούτω καθεξής. Ε, εγώ νομίζω ότι το μόνο που αληθεύει είναι ότι δεν είναι έτοιμη ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε όχι νωρίτερα από τον Απρίλιο. Πολύ φοβάμαι ότι μετά τον Απρίλιο ε, θα απουσιάζετε κι εσείς πνευματικά από τις Βρυξέλλες, ε, όσο και εμείς, διότι κι εσείς πλησιάζετε το τέλος της θητείας σας. και πολύ φοβάμαι ότι υπό την εμπνευσμένη ηγεσία του Προέδρου Μπαρόζο και δεδομένου του κλίματος που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να προσδοκούμε οποιαδήποτε πρόταση από πλευράς αυτής της Επιτροπής και δεν πρόκειται μόνο για την οδηγία ποιότητας καυσίμων στην Ευρώπη. Είναι ένα μήνυμα που περνάμε ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Οι ασφαλτούχοι είναι τα, τα πιο ε, τα χειρότερα ορυκτά καύσιμα ως προς τη ρήπανση που έχουμε και όχι μόνο αυτό, ε, δημιουργούν ένα πελώριο πρόβλημα βιοπικιλότητας. Έχουμε και το Καζακστάν, τη Ρωσία και την Ιγυρία πέρα από τον Καναδά. στην Νιγηρία απειλούνται ακόμη τα παρθένα δάση που έχει. Θα εξακολουθεί να έχει προς το παρόν. Εάν λοιπόν δεν ε, ε, εγκρίνουμε μια φιλόδοξη οδηγία, τι μήνυμα περνάμε στον υπόλοιπο κόσμο. Παρακαλούμε, συνεχίστε ε, αυτά που κάνετε με την ασφαλτούχο άμμο. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Καναδάς, είναι και η Ρωσία, είναι και το Καζακστάν, είναι και η Νιγηρία. Είναι εσφαλμένο αυτό το μήνυμα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Για ώρες θα μπορούσα να σας μιλάω ε, και να μου ε, αντιλέγετε εσείς, αλλά δυστυχώς ε, Η ομοία αλήθεια είναι ότι ο Επίτροπός σας δεν καταφέρει να προωθήσει την πρόταση στο σώμα των Επιτρόπων και ο Επίτροπος Ποτόσνικ το ίδιο πρόβλημα είχε με το σχιστολιθικό και άλλα συναφή και με τις πλαστικές σακούλες που μόλις συζητήσαμε επίσης. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Έχουμε μια ομάδα 50 διακεκριμένων επιστημόνων που ε, απέστειλαν ε, γράμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια σειρά επιχειρημάτων ε, σχετικά με το, ε, τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προωθήσουμε την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, ε, για, συγκεκριμένα για την ασφαλτούχο άμμο. Ε, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, απαντήσει, να δημοσιοποιήσει την απάντηση προς αυτή την επιστολή, διότι αξίζει το κοινό έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο για αυτό το ζήτημα δεδομένων των επιπτώσεων της ασφαλτού άμμου τόσο επί της βιοποικιλότητας όσο και επί του περιβάλλοντος. Ε, Μπάς Έιχουτ, ε, ευχαριστώ. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, μπορείτε να μου εξηγήσετε παρακαλώ γιατί δεν ε, υπάρχει καμία συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ το συνολικό πακέτο, παραδείγματο χάρη, υπαναχωρείται από τη στοχοθέτηση για τι ανανεώσιμες ε, και ε, δίνεται μεγαλύτερη σημασία τώρα πλέον στου στόχου για τη μείωση των εκπομπών των φλουαρίων θερμοκηπίου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολουθεί την ίδια λογική στον τομέα των μεταφορών, διότι αυτό θα σήμαινε ότι η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων έχει ακόμη περισσότερη σημασία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή δεν το κάνει αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει μια ανησυχία ε, ότι λόγω του πακέτου 2030 όπου ε, ε, έχει παγιδευτεί η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, δεν θα αναλυφθεί πλέον καμία δράση σε αυτό το τομέα. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν αληθεύει αυτό και ότι ε, Φέτο κατά την τωρινή θητεία θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μία πρόταση ε, για την ποιότητα του καυσίμων τουλάχιστον μέχρι το 2020 και βλέπουμε μετά μέχρι το 30. Σας ευχαριστώ και κλείνοντας θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το την επιστολή από τους ε, επιστήμονες και για την συνάντηση με τους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρκετούς εκπροσώπους. Δεν ε, θεωρώ ότι είναι πρόβλημα να διαθέσουμε το γράμμα αυτό, την ε, επιστολή αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει ζητηθεί πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να το χορηγήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο ερώτημα είναι ενδεχομένω του Μπασάικατ είναι λίγο πιο δύσκολο να απαντηθεί με απλό τρόπο. Νομίζω καταρχάς ότι θα υπάρξει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη να προσμετρούνται οι εκπομπές από τα καύσιμα αν έχουμε θέσει το στόχο του 40% σε όλη την οικονομία. Κάποιο από αυτό το ποσοστό θα προέλθει από το σύστημα εμπορία ρήπων, λοιπόν, κάποιο άλλο όχι. Θα υπάρξει απόφαση λοιπόν για την κατανομή και την, ε, το διαμοιρασμό των προσπαθειών για να πετύχουμε τον στόχο του 40% θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να συλλεχθούν πληροφορίες για τα καύσιμα που ε, υπησέρχονται στον τομέα των μεταφορών, το 20-25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και θεωρώ ότι υπάρχει νόημα να υπάρχει μια μεθοδολογία για να ε, τα ορυκτά κάψιμα και σε ό,τι αφορά και τα βιοκάψιμα θα πρέπει να υπάρχει αξιόπιστη μεθοδολογία και για τα αρκτά καύσιμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι η για ότι η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων θα ε, πάυσει να ισχύει από το 2020 και μετά. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Και επίσης δεν νομίζω ότι στέκει το ότι δεν υπάρχει κανένα στόχος για τις μεταφορές ε, η Λευκή Βίβλο για, το, για την ε, για τις μεταφορές περιλαμβάνει ένα στόχο το 2050, το οποίο είναι ο στόχος. Αλλά στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής συζητάμε το στόχο του 2030 και του 2050 για τις μεταφορές. για τα εφαρμοστικά μέτρα για το 7α. Ε, είμαστε, έχουμε καθυστερήσει. Ναι, ασφαλώς και έχουμε καθυστερήσει. Μπορεί οι κοινικοί να μας πούν ότι δεν χρειάζεται μέχρι το 2020, γιατί αυτό είναι ο στόχος μέτρησης, άρα δεν έχουν χαθεί τα πάντα. Και θέλουμε να υποβάλουμε την πρόταση αυτή. Είμαι πεπισμένος, γι' αυτό το ίδιο και ο Επιτροπός μου. Μπορεί να λέτε ότι έχει ολοκληρωθεί η θητεία σχεδόν όλου του κόσμου αλλά θεωρώ ότι συμφέρει όλους μας να προωθηθεί το θέμα αυτό και την ε, Παρασκευή το απόγευμα έχω μία συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα για να προωθήσω και να συζητήσω το θέμα αυτό. Άρα όλους μας συμφέρει και όλοι τον προωθούμε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος, κοιτώντας και προς τους συναδέλφους. δεν δεν θέλει κανείς άλλος ε, το λόγο. Να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους μου λοιπόν που συμμετείχαν στην ε, συζήτηση. Ολοκληρώσαμε έτσι την ημερησία διάταξη. Αύριο στις 10 συνεχίζουμε εδώ στη συζήτησή μας και από τις 9 έως τις 10 θα συνεδριάσουμε και κλεισμένων των θυρών ε, οι συντονιστές. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.